Colleagues, good afternoon. Uh, Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, σας ε, καλωσορίζουμε ως πρόεδρος της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, υποψήφιο τον προτινόμενο επίτροπο, κύριο Μπρετόν, και επίσης ε, και το μέλο της Επιτροπής Έρευνας και Ενέργειας θα συμπροεδρεύσουμε και βεβαίως θα ήθελα να καλωσορίσω και τα μέλη της ΙΜΚΟ και της ΙΤΡΕ ε, γιατί η συνεδρίαση αυτή ε, διεξάγεται από κοινού. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, παρακαλέσω να καθίσετε και ας ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της Γιούρη και της ΚΑΛΤ. Βλέπω ότι είσαστε κοντά μας, είναι οι πρόεδροι αυτών των δύο επιτροπών. Οι επιτροπές έχουν σχέση με την ακρόση και έχουμε προσκαλέσει και την Επιτροπή Μεταφορών και την Υποεπιτροπή ΣΕΝΤΕ. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω υπενθυμίζοντάς σας ότι η ακρόαση αυτή κατά κύριο λόγο έχει ως στόχο να επιτρέψει στα μέλη και των δύο επιτροπών να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις. Πρώτον, κατά πόσον ο προτινόμενος επίτροπος ε, έχει τα απαραίτητα προσόντα για να ενταχθεί στο σώμα των ε, επιτρόπων και δεύτερον, κατά πόσον έχει τα προσόντα για να επιτελέσει τα καθήκοντα που θα το ανατεθούν. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή ΙΜΚΟ είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της κοινή αγοράς συμπεριλαμβανομένων μέτρων που έχουν σχέση με τον εντοπισμό και την άρση εμποδίων για την ολοκλήρωση της κοινής αγοράς ε, ε, την προστασία των οικονομικών ε, συμφερόντων των καταναλωτών. Είναι επίση αρμόδια για θέματα πολιτική και νομοθεσία που σχετίζονται με την εφαρμογή των κανόνων τη κοινή αγορά και τα δικαιώματα των ε, καταναλωτών. Γνωρίζετε επίση πολύ καλά ότι η Επιτροπή μας προσβλέπει σε αυτήν την ακρόση για να κατανοήσει την προσέγγιση του κ. Μπετρών σε σχέση με τα θέματα που προανέφερα. Επιθυμούμε να γνωρίζουμε πώς ο προτινόμενο Επίτροπος προτίθεται να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα και τι είδους ενέργειες προτίθεται να προτείνει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η κοινή αγορά για υπηρεσίες και αγαθά είναι καθοριστική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καθοριστική για την επιβίωση των επιχειρήσεων, είναι κλειδί ε, κατ' ουσίαν και για το ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα κατά νου την επιτυχία της κοινή αγοράς και το γεγονός ότι προφανώς και εξαρτάται από τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έγκαιρη εφαρμογή αυτών των κανόνων είναι καθοριστική σημασία για να εκμεταλλευτούμε πλήρω τι δυνατότητε που προσφέρει η κοινή αγορά. Και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να ενισχύουμε και να εμβαθαίνουμε την κοινή αγορά, περιορίζοντα εμπόδια ε, για τα ε, προϊόντα και για της τις να καταπολεμήσουμε την ε, κατάτμιση της αγοράς και επίσης να αποφύγουμε και τεχνητούς, ε, τεχνητές διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις νέες αγορές και τις ψηφιακές αγορές γιατί θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι καθοριστική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και για τη βελτίωση των ε, υπηρεσιών και των προϊόντων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο τομέας των υπηρεσιών είναι καθοριστική σημασία για την ευημερία, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και για την ευημερία των καταναλωτών σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά. Αυτό λοιπόν που καλούμεθα είναι να εφαρμόζουμε τους κανόνες, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία μας ενδείκνυται σε αυτή την ψηφιακή εποχή και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, της τεχνικής πρόοδου, ε, να διασφαλίσουμε, να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι ο προτινόμενος ε, Επίτροπος θα κατανοήσει όλες αυτές τις ανησυχίες μας για το μέλλον και το πόσο σημαντικό είναι να εστιάσει κανείς την εύρυθμη λειτουργία έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την προσαρμογή στη σύγχρονη οικονομία. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ε, που μου δίνεται η δυνατότητα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο ε, Κονζδεύσκη από την Επιτροπή ΕΜΚΟ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τεσάταρ. Καλωσορίζω όλα τα μέλη από όλε τι επιτροπέ που συμμετέχουν σε αυτή την κοινή ακρόαση και ειδικότερα τον υποψήφιο επιτρόπο κύριο Τιρή Μπρετό. Όπως πάντα η ακροασή μα μεταδίδεται ζωντανά στην ιστοσελίδα μας. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να καλωσορίσω και όλους όσοι μας παρακολουθούν από τη μαγνητοσκόπηση. Να υπενθυμίσω ότι η ΙΤΡΕ είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για τη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τις νέες τεχνολογίες, ε, το διάστημα, την κοινωνία των πληροφοριών, την τεχνολογία πληροφοριών και τα δίκτυα επικοινωνιών και τις υπηρεσίες. Η ακρόαση αυτή είναι πολύ σημαντική για την Ήτρε δεδομένου ότι το χαρτοφυλάκιο της εσωτερικής αγοράς περιλαμβάνει την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την αμυντική βιομηχανία και το διάστημα. Όλοι αυτοί οι τομεί θα παίξουν κρίσιμο ρόλο για την περαιτέρω εξέλιξη τη Ένωση σε αυτή τη θητεία και την επόμενη. Να σας εξηγήσω τώρα πώς ε, θα διεξαχθεί η σημερινή ακρόαση. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες ε, οδηγίες, ε, ο υποψήφιος Επιτρόπος θα αξιολογηθεί βάσει των γενικών του ικανοτήτων, της ευρωπαϊκής δέσμευσης και της προσωπικής ανεξαρτησίας. Θα αξιολογηθεί επίσης, θα αξιολογηθούν οι γνώσεις ε, για τα σχετικά χαρτοφυλάκια και οι ικανότητες επικοινωνίας. Πριν από την ακρόαση, ο υποψήφιος επίτροπος απάντησε γραπτός σε ένα προπαρασκευαστικό ερωτηματολόγιο. Οι γραπτές απαντήσεις έχουν διανεμηθεί στα μέλη σε όλες τις γλώσσες. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων δεν έχει θέσει καμία ένσταση στη διεξαγωγή της ακρόασης. Η συζήτηση θα δομηθεί ω εξή. Ο κύριος Μπρετόν θα κληθεί να κάνει μια εναρκτήρια ε, δήλωση, όχι μεγαλύτερη των 15 λεπτών, θα είμαστε πολύ αυστηροί με το χρόνο. Στη συνέχεια, στο τέλος της ε, ε, συνεδρίασης θα έχει και άλλα 5 λεπτά για την τελική του παρουσίαση. Μετά από την εισαγωγή θα υπάρχει χρόνος για 25 ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές και η συζήτηση θα γίνει σύμφωνα με χρονοθυρίδες 5 λεπτών για τον καθένα, ένα λεπτό για τρία λεπτά για τις ερωτήσεις και 2 λεπτά για τις απαντήσεις από τον κύριο Μπρετών. Σε περίπτωση επερωτήσεων, οι ερωτήσεις δεν πρέπει να διαρκούν περισσότερο από ένα λεπτό, με ένα λεπτό για την απάντηση. Να σας υπενθυμίσω ότι οι επερωτήσεις θα πρέπει φυσικά να γίνονται από το ίδιο μέλη και να σχετίζονται με την αρχική ερώτηση. Ο πρώτος γύρος των 7 ερωτήσεων θα γίνει από του εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων. Ο δεύτερο γύρο των 18 ερωτήσεων βασίζεται στη συνολική κατανομή των ερωτήσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων των μη εγγεγραμμένων. Η διερμηνία θα παρέχεται σε 23 γλώσσες. Έτσι λοιπόν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δική σας γλώσσα, αλλά παρακαλώ να θυμάστε μην μιλάτε υπερβολικά γρήγορα για να μπορεί να διεξαχθεί σωστά η διερμηνία. Τώρα σας δίνω το λόγο στον υποψήφιο επίτροπο για την εναρκτήρια δήλωσή του που όπως είπα δεν πρέπει να διερκέσει πάνω από 15 λεπτά. Παρακαλώ κύριε Μπρετό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Θα αρχίσω εκφράζοντας τον απόλυτο σεβασμό μου για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σας ε, ευχαριστήσω όλους γι' αυτό, για ό,τι κάνετε κάθε μέρα στην υπηρεσία της Ευρώπης και των Ευρωπαίων πολιτών. Πρώτα απ' όλα όμως επιτρέψτε μου να παρουσιάσω τον εαυτό μου, γιατί ξέρω ότι μέσα από εσά θα αποκτήσω την νομιμότητα να δράσω ως Επίτροπος στη συνέχεια. Ας μπούμε λοιπόν ε, στην ουσία του θέματος. Πρόκειται για το εξής. Εγώ είμαι παππούς. Πολύ ευτυχής παππούς ε, του Λουί και της Άβα που είναι γερμανάκια, τα εγγονάκια μου και ζουν στο Βερολίνο. Ε, Πολλοί ισχυρίζονται ότι ε, έχω μια ωραία ζωή και εγώ όπως και πολλοί άλλοι έχω πράγματι μια πολύ ωραία ζωή και θα ήθελα να πω το light motif της ζωής μου είναι το πάθος. Αυτό είναι το οδηγό νήμα που με καθοδηγεί. Το πάθος των επιστημών και της τεχνολογίας πρώτα απ' όλα που πάντα τροφοδότησαν τον προβληματισμό μου προκειμένου να προλάβω αλλαγές και να προσπαθήσω να τις καταλάβω όσον αφορά το περιβάλλον, τον κοινωνικό χώρο, τον κόσμο μας γενικότερα. Έπειτα το πάθος της νεότητας για να μεταφέρει μηνύματα, να επικοινωνήσει, να διδάξει, της οικονομίας, την επιχειρήσω, θα έλεγα μάλιστα το επιχειρηματικό πνεύμα, το επιχειρίζεστε. Επίσης το πάθος για το δημόσιο χώρο, για να υπηρετήσω, να συνεισφέρω ε, παντού και όλους όσοι εργάζονται για το δημόσιο συμφέρον. Το πάθος επίσης για την Ευρώπη μας, για την ιστορία της, για τις αξίες της και για την ποικιλομορφία της. Είμαι φτιαγμένο από όλα αυτά τα πάθη και σήμερα μου προσφέρετε, εφόσον εσείς το δεχτείτε, η δυνατότητα να βάλω όλη μου την ενέργεια και να συνεργαστώ μαζί σας με ένα όραμα και μία φιλοδοξία για την Ήπειρό μα μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος περνάει άνευ προηγουμένου ανατροπές. Και αυτές οι ανατροπές, αυτές οι αλλαγέ, η εκλεγμένη πρόεδρο Φοντερ Λάιεν τις έχει περιγράψει πάρα πολύ καλά. Είναι η κλιματική αλλαγή, είναι η ψηφιακή αλλαγή, αλλά είναι επίση και οι νέε γεωπολιτικέ τάσει που είναι άνευ προηγουμένου αυτόν τον αιώνα. Και επίσης αυτό που κάνει τόσο άνευ την σημερινή κατάσταση για όλους μας είναι ότι συγχρόνως όλες αυτές οι προκλήσεις συσσωρεύονται την ίδια στιγμή στην Ήπειρό μας. Κυρίες και κύριοι προβουλευτές, Μίλησα για το πάθος μου, για τη δέσμευσή μου υπέρ της Ευρώπης, όπως ισχύει και για σας. Και πάντα ήμουν ένας πεπισμένος Ευρωπαίος σε όλα τα στάδια της ζωής μου. Από τότε που νέος έφτιαξα μια πρώτη επιχείρηση, στη συνέχεια όταν έγινα ερετός, στη συνέχεια ε, υπουργό και μετά ειδικό για τις τεχνολογίες ε, των πληροφοριών. Η εντολή σας, εφόσον φυσικά με εμπιστευτείτε, εγγράφεται πλήρως σε αυτήν ακριβώς τη δέσμευση. Θα είμαι ευθύ μαζί σα. Επίγει να ετοιμάσουμε την αυριανή ανάπτυξη επενδύοντα ήδη από σήμερα στι βασικέ τεχνολογίε για το μέλλον. Για παράδειγμα, το PG, αλλά πρέπει ήδη να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για το 6G, για την τεχνητή νοημοσύνη, το νεφο, αλλά και τι θα γίνει μετά το νεφο, για την πληροφορική αιχμή, για το διαδίκτυο των πραγμάτων, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, blockchain. Και έπειτα, δεν θα σα εκπλήσει, τουλάχιστον όσους με γνωρίζετε, με ενδιαφέρει η κβαντική τεχνολογία. Όλες αυτές οι τεχνολογίες είναι τεχνολογίες που πρέπει να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε, να γνωρίζουμε καλά και να μπορέσουμε όσο μεγάλη βιομηχανική δύναμη στον κόσμο να δράσουμε. Ακριβώς αυτό το αντικείμενο του χαρτοφυλακίου μου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι προκλήσει για την αυριανή ανάπτυξη και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κατανοήσουμε τον ψηφιακό χώρο, ο οποίος έχει να κάνει με όλες τις διαστάσεις της εσωτερικής αγοράς, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Πρόκειται για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, πρόκειται για τη βιομηχανία 4.0, πρόκειται για όλες τις υπηρεσίες, το πολιτιστικό κλάδο, ε, το περιεχόμενο, ε, προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την άμυνα, με τους ηλεκτρονικούς ε, πολέμους, αλλά ακόμα και με το ίδιο το διάστημα και τις τεχνολογίες του. Πρόκληση λοιπόν για μας είναι να οργανώσουμε, να ρυθμίσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες, τεχνολογικές, βιομηχανικές, πολιτιστικές, σε αυτόν τον χώρο που σήμερα είναι ένας χώρος πληροφορίας και με ελεύθερη πρόσβαση και ισότιμη κατανομή, όπως το έχουμε ήδη κάνει τον προηγούμενο αιώνα για τους άλλους τρεις χρόνους που διαμόρφωσαν την ανθρώπινη δραστηριότητα που είχε να κάνει με το έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα τέταρτο χώρο, ο οποίος μπαίνει πάνω από τους τρεις προηγούμενους, χωρίς όμως αποκλεισμού και πρόκειται για τον χώρο της πληροφορίας. Και γι' αυτόν χρειαζόμαστε ένα ισότιμο πεδίο δράσης, όπως και για τους άλλους τρεις. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν η φιλοδοξία μου για το χαρτοφυλλόκιό μου θα το ορίσω ως εξής. Προστασία, ε, αλλαγή και προβολή στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει προστασία για να προστατεύουμε την εσωτερική μας αγορά και τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Αυτή η προστασία τη εσωτερική αγορά ισχύει επίση και για του ευρωπαίου εργαζόμενου, οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να προσφέρουν τι υπηρεσίε του σε όλε τι χώρε μέλη τη Ένωση, έχοντα την εγγύηση ότι αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά του προσόντα. Έπειτα βέβαια, οι κανόνε τη εσωτερική αγορά πρέπει να τηρούνται σωστά, γιατί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα σύγκληση και ανάπτυξη για όλε τι χώρε τη Ένωση. Και επιμένω, για όλου. Και σε αυτό είμαι αδιάλακτο για την προστασία των εργαζόμενων και τι συνθήκε εργασία του. Επίση, θα φροντίσω στη εσωτερική μα αγορά να μα προστατεύει από τον εξωτερικό ανταγωνισμό όταν αυτό είναι αθέμητο. Πρέπει να κινητοποιούμεθα χωρί να είμαστε αφελεί, ώστε να πετυχαίνουμε ε, πιο δίκαιο εμπόριο παντού στον κόσμο. Και αυτά βέβαια σε συνεργασία με τον Φιλ Χόγκαν. Ο ρόλο μου επίση θα είναι να προστατεύω τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, τι startup, να συνοδεύω τι νέε μορφέ απασχόληση, ε, φροντίζοντα να υπάρχει ισότιμο ανταγωνισμό με του γίγαντε τη υπήρου μα. Και επίση φροντίζοντα παντού να σεβόμαστε τα κοινωνικά δικαιώματα. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο, την ε, τροποποίηση, την αλλαγή, την προσαρμογή, γιατί πρέπει με φιλόδοξε βιομηχανικές πολιτικές να συνοδεύσουμε τις αλλαγέ που λαμβάνουν χώρα ώστε να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας και να τις καταστήσουμε πιο ανταγωνιστικές. Και εδώ μιλάμε και για τις αλυσίδες αξιών. Πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας, είναι πολύ βασικό για μένα, το έχω ήδη πει, η κοινωνική μας ευθύνη σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει μαζί να φροντίσουμε οι αλλαγές αυτές να είναι αλλαγές από τις οποίες όλοι να μπορούν να αποφεληθούν παντού στην Ευρώπη. Στον όλο αυτό το συνοδευτικό που αναλαμβάνω εγώ, η προτεραιότητά μου είναι σαφής. Δεν θα αφήσω κανένα στα μισά του δρόμου. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό ε, Κυρίω μέσω της κατάρτισης και αυτό θα το κάνω σε συνεργασία με τον Βάλτη Ντομπρόφσκι και τον φίλο μου Νικόλα Σμιτ. Για μένα θα είναι μεγάλο μου μέλημα. Όλες αυτές οι αλλαγέ ψηφιακέ, οικολογικέ κτλ. ξέρω θα δημιουργήσουν σημαντικές αλλαγέ για πολλούς από τους συμπολίτε μας και καταλαβαίνω τον φόβο απέναντι στην τεχνολογία αλλά εδώ πρέπει να προλάβουμε, να συνοδεύσουμε τον κόσμο σε αυτές τις αλλαγές, κάτι που αποτελεί ευκαιρία, έτσι ώστε όλοι όσοι χρειάζονται νέα κατάρτιση να μπορέσουν να την αποκτήσουν για να βρουν μια καινούργια δουλειά. Για μένα αυτή είναι η τρίτη πρόκληση και αυτό ακριβώ συμπεριλαμβάνω στο και ο εξίσου όπως και τα προηγούμενα. Πρόκειται για την οικολογική και την ψηφιακή πρόκληση. Εδώ θέλω να πω επίσης ότι πρέπει να στηρίξουμε μια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η εσωτερική αγορά πρέπει να έχει κανόνες που να ευνούν όλες τις επιχειρήσεις, όλες επιμένω, μικρές, μεσαίες, μεγάλες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι νέοι κανόνε ανταγωνισμού είναι συμβατοί με μια σύγχρονη οικονομία και συνεισφέρουν στο να αναδυθεί μια νέα ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανία και στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο το Θύμισε αυτό εξάλλου και εκλεγμένη πρόεδρος Φοντερ Λάιν. Επίσης θα συνεργαστώ με όλο το Σώμα των Επιτρόπων, με την ε, Μαργαρίτα Φεστάγκερ για να συνεισφέρω από τη δική μου τη θέση για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική η οποία να συμπεριλαμβάνει τις νέες αυτές προκλήσεις και κυρίως πρέπει να αναρωτιόμαστε χωρίς ταμπού. Τα ψηφιακά και ο συσχετισμός δυνάμεων πώς αλλάζει στον κόσμο και πώς πρέπει να προσαρμόζονται όλες οι ευρωπαϊκές πολιτικές, όλες. Γιατί στόχος μας πρέπει να είναι να δημιουργούμε στρατηγικές για κάθε κλάδο και αλυσίδες αξιών παντού. Είτε πρόκειται για τη βιομηχανία, είτε πρόκειται για τι υπηρεσίε και στις υπηρεσίε, Να λάβουν υπόψη μα το έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με τον τουρισμό, γιατί εδώ υπάρχουν αλλαγές και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις αλλαγές των οικοσύστημάτων όταν μιλάμε για τουρισμό και η Ευρώπη πρέπει να διατηρηθεί σαν ε, πρώτος προορισμός τουριστικός στον κόσμο. Επίσης, σκέφτομαι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τον πνεύμονα της οικονομίας μας, αλλά και τη startup. Πρέπει να τις βοηθήσουμε να προσαρμόζονται, αλλά να τους διευκολύνουμε και τη ζωή με κάθε μέσο, για να μπορούν να διασφαλίσουν με τη σειρά τους στην εσωτερική αγορά ε, την εύκολη πρόσβαση πρέπει να έχουν οι ίδιες εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση στις δημόσιες αγορές. Έπειτα, έρχομαι στο τρίτο, προστασία. Και αυτό είναι το τρίτο, τρίτος μου άξονας. Η εσωτερική αγορά είναι ένα βήμα το οποίο επιτρέπει να προχωρήσει στην τεχνολογική της κυριαρχία η Ευρώπη και τη βιομηχανική και την πολιτιστική και να προβληθεί στον κόσμο. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε να το φροντίσουμε για τον ήπειρό μας και να μην ξεχνάμε βέβαια ποτέ τις επιπτώσεις στην κοινωνία που μπορεί να έχει οποιαδήποτε πολιτιστική πολιτική. Η παραγωγή βίντεο, για παράδειγμα, ε, περνάει από μια έκρηξη. Τι συνέπειες έχει αυτό. Η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να μην συντονίζεται. Και αυτό θα φροντίσω και εγώ να το κάνω με την ε, κυρία Φερχέγεν, που είναι η επίτροπος, η αρμόδια για τα πολιτιστικά. Θα συνεργαζόμαστε λοιπόν και δεν θα υπάρχει κατακαιρματισμός με ένα συγκεκριμένο σχέδιο υπό την Μαρία Καμπριέλ. Γιατί για μένα η πολιτιστική διάσταση και για την Ήπειρό μα και τον μόνο σας το πω εδώ, έχει εξίσου σημασία όπως και η οικονομική μας άνθηση. Εδώ λοιπόν, εκτός από τη τεχνολογική κυριαρχία, θέλω να μιλήσω και για τη στρατηγική μας. Η προβολή μας σημαίνει και σημαντικές επενδύσεις στις μελλοντικέ τεχνολογίες, στα ψηφιακά, στα ε, οχήματα που θα οδηγούνται μόνα τους, στις ηλεκτρικές ε, μπαταρίες, ε, το υδρογόνο κλπ. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται βέβαια στην ψηφιακή πράξη για να ρυθμιστούν όλες αυτές οι μεγάλες ψηφιακές προκλάσεις. Πρέπει να γίνουμε λοιπόν και εμείς ε, με συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κανόνες και να προχωρήσουμε έτσι. Εμείς ακολουθούμε και τον δρόμο της κυρίας Φαστάγκερ για ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό για την τεχνητή νοημοσύνη με εθικές τυχές, αλλά και τεχνολογικές. Και αυτό θα φροντίσω να το κάνω και για το διάστημα. Η Ευρώπη πρέπει βεβαίως να συνεχίσει να είναι αυτόνομη όσον αφορά το διάστημα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση για το Κοπέρνικους και το Γκαλέιο. Μαζί με την Μαρία Γκάπριελ ε, επιταχύνουμε την ανάπτυξη για ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία. Σε όλα αυτά, η άμυνα φυσικά θα αποτελέσει μια σημαντική διάσταση, γιατί τελικά υπάρχει αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο θα πρέπει να βοηθήσει όλες ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έπειτα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό και το γνωρίζετε και σκοπεύω προσωπικά σε αυτό να το λάβω υπόψη μου σε όλες τις διαστάσεις του χαρτοφυλακίου μου. Για όλη την εσωτερική αγορά, από τη μία άκρη στην άλλη. Γιατί είναι διαφορετική σημασία. Έπειτα, <clears throat> πρέπει να κινητοποιηθεί ο καθένας μας για την καταπολέμηση της ε, θέρμανσης του πλανήτη. Έτσι λοιπόν, σε συνεργασία με τους συναδέρφους μου, θα προχωρήσω κι εγώ στην περίφημη πράσινη συμφωνία με φιλοδοξία. Επίσης, θα βοηθήσω και ε, μαζί με τον Φρανς Τίμερμενς και ό,τι έχει να κάνει με το Green Deal γύρω από μια στρατηγική για την κυκλική οικονομία και για να, επαν, προσανατολιστεί η πολιτική μας. Θα συνεργαστώ μαζί σας στενά. Θα είμαι πάντα εδώ για να σας ακούω και για να δείχνω τη θέλησή μου, γιατί την έχω. Είναι μια βούληση για όλα τα στάδια οικοδόμησης της Ευρώπης υπέρ του μέλλοντός μας και υπέρ της Ευρώπης και με όλους, όλες τις πλευρές. Πρέπει να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις, τα σωματεία, τους κατανοητές, τα συνδικάτα, όλοι έχουν ένα λόγο και εγώ θα τους ακούω όλους, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές. Όταν έχουμε πολλές ζωές μέσα σε μια ζωή και βρισκόμαστε εδώ ενώπιόν σας σήμερα, σημαίνει ότι το θέμα της ηθικής και της σύγκρουσης συμφερόντων είναι κάτι που μας απασχολεί βαθιά. Και γι' αυτό το συγκεκριμένο θα μιλήσω χωρίς περιστροφές. Δεν υπάρχουν πολλές λύσεις. Εγώ είμαι ριζοσπάστης, το λέω ριζοσπάστης. Πάντα με ενδιαφέρει το κοινό συμφέρον. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Και έτσι λοιπόν βρίσκομαι εδώ σήμερα μπροστά σα. Χωρί να έχω κανένα συμφέρον οικονομικό σε καμία επιχείρηση και αυτό το λέω έχω πουλήσει όλε μου τι μετοχέ πριν καν έρθω εδώ και έχω παραιτηθεί από όλε μου τι εντολέ αλλά αυτοί που πιστεύουν ότι επειδή έχω αναλάβει στο παρελθόν κάποιες ε, αρμοδιότητες στις επιχειρήσεις μπορεί να τι ευνοήσω κάποια στιγμή. Και γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει, γιατί υπάρχουν κανόνε εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιο συγκεκριμένα τα άρθρα 2, 6 και 4 του κώδικα διοντολογία των επιτρόπων. Και έτσι όπω και όλοι οι υπόλοιποι οι επίτροποι, έτσι και εγώ θα φροντίσω τα άρθρα αυτά να τα σέβομαι απόλυτα με κάθε διαφάνεια. Όπω προβλέπετε λοιπόν στον ε, κώδικα διοντολογία, αν υπάρξει θέμα οικονομικού συμφέροντο ή οτιδήποτε άλλο, εγώ θα κοινοποιήσω αμέσω στην Πρόεδρο. Αυτά λέει ο κώδικας διοντολογίας. Και αν με βεβαιώσετε στη θέση του Επιτρόπου, θα κάνω το ίδια και σε αυτή την υπόθεση και από αυτή τη θέση, όπως έκανα και με αδιαλαξία και με αυστηρότητα όταν έγινε υπουργό Οικονομίας στη Γαλλία. Αν βεβαιώσετε τη θέση μου, σας το λέω δυνατά και το βροτοφωνάζω. Ένα πράγμα θα μου απασχολεί πάντα, το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Και αυτή θα είναι η πηξίδα μου. Σας ευχαριστώ. Ε, thank you. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα ήθελα να καλέσω τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων για τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. ΕΛΚΑ, ο κύριο Φρανσουά Ξεβιέ Μπελάμι, παρακαλώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, η αποστολή που σας αναμένει είναι καθοριστική για το μέλλον μας. Για πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι δεν αντιλήφθηκε την έκταση της παγκοσμιοποίησης. Φτιάχναμε κανόνες αντί για στρατηγική και μερικές φορές θέσαμε τις βιομηχανίες μας σε εύθραυστη θέση αντί να υποστηρίζουμε. Σε ορισμένους κλάδους βιομηχανικούς οι επιχειρήσεις βρέθηκαν σε ανταγωνισμό με συναγωνιστές που δεν τηρούν κανένα κανόνα από αυτούς που έχουμε στην Ευρώπη και που συχνά έχουν τεράστια υποστήριξη από τα κράτη τους. Έτσι χάσαμε πάρα πολλέ βιομηχανικές μάχες, θέσεις απασχόλησης και τεχνογνωσία. Η κρίση που ζούμε αυτή τη στιγμή μα αναγκάζει να εγκαταλείψουμε την αφέλεια. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει για να εξισορροπήσει την παγκοσμιοποίηση. Επιβάλλεται οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά και οικολογικά. Πώ προβλέπετε ε, την αλλαγή που μα αναμένει. Τι προτεραιότητες ε, θα υιοθετήσετε για να δώσουμε οξυγόνο στι επιχειρήσει τη χώρα μα και στις οικονομίε μα. Θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο να επενδύσουμε σε στρατηγικές ε, αλυσίδες αξιών που υφίστανται ιδιαίτερα, ε, ιδιαίτερο ανταγωνισμό χωρίς καμία απολύτως ισορροπία. Ευχαριστούμε κύριε Μπελαμή για αυτή την ερώτηση. με απασχολεί στο επίκεντρο της ε, πολιτικής που θα αναλάβω στο χαρτοφυλακείο μου και έχετε δίκιο, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς. Τώρα πρέπει να αποφασιστούν όλα. Έτσι θα εστιαστώ σε τρει μεγάλε προτεραιότητε. Πρώτα απ' όλα τον εξυγχρονισμό τη ενιαία αγορά. Υπάρχουν ακόμα πολλά να γίνουν, το γνωρίζουμε. Χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα. Πρέπει φυσικά να χαμηλώσουμε τα σύνορα. Ε, θα το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια τη ακρόαση. Επίση, κάτι καθοριστικό σε αυτό το χαρτοφυλάκιο θα είναι ότι θα πρέπει να δράσουμε έτσι ώστε όλοι οι κλάδοι των οικονομιών μας, οι υπηρεσίες, η βιομηχανία, 99,8% μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μάλιστα είναι η βιομηχανία μας μετά, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, όλα χαρακτηρίζονται από τις ψηφιακές τεχνολογίες, οπότε ο ρόλος μου θα είναι να δράσω παντού για να βοηθήσω το σύνολο των κλάδων να μετασχηματιστούν. Αλλά έχετε δίκιο, χρειάζονται και μεγάλοι όμιλοι, οι οποίοι να μπορούν να αγωνιστούν εισάξια με τους κολοσσούς ε, εκτός Ευρώπης και συχνά εκτό Ευρώπη δεν έχουν του ίδιου κανόνε ε, όπω έχουμε εμεί το είπατε και γι' αυτό θα ενθαρρύνουμε τι στρατηγικέ μεγάλων αλυσίδων όπω είπατε, το υπενθυμίζω. και οι τεχνολογίε κλειδί είναι βασικέ, θα πρέπει να επενδύσουμε μαζικά σε αυτέ. Ε, θα αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη την διανοητική ιδιοκτησία την βιομηχανία, την ασφάλεια στον χώρο, διότι αυτό το τελευταίο θα παίξει σημαντικό ρόλο. Το σύνολο του χαρτοφυλακίου πιστεύω ότι αποκρίνεται απόλυτα και μας παρέχει τα μέσα να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μόλις αναφέρατε. Yeah, follow up question, please, Mr. Επερώτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, για την απάντησή σας. Αναφέρατε ακριβώς ε, μεταξύ των διαφόρων κλάδων κάποιους που έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα, διότι αποτελούν προϋπόθεση για το μέλλον μας, όχι μόνο οικονομικά, αλλά θα καθορίσουν και την πολιτική μας αυτονομία. Τα θέματα ασφάλειας, για παράδειγμα, η αμυντική βιομηχανία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το οποίο γνωρίζετε καλά. Αυτό το υποστήριξε στην τελευταία του θητεία το Κοινοβούλιο μέσω ενός εργαλείου συλλογικών επενδύσεων. Τι θεωρείτε ότι θα γίνει για το μέλλον. Ε, σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να αποκτήσει στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη σε βιομηχανικό επίπεδο. Και τώρα, όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ποιε δράσει θεωρείτε ότι πρέπει να έχουν προτεραιότητα για να καλύψουμε τι καθυστερήσει. Ποιε είναι ε, οι φάσει που θεωρείτε ότι πρέπει να διέλθουμε για να διασφαλίσουμε την ε, προστασία των πολιτών και των κρατών μα Επ' αυτού του θέματο, δεν είναι μόνο η δική μα οικονομική επιβίωση που διακυβεύεται, αλλά και το μέλλον των ελευθεριών και τη δημοκρατία μα πολύ ευρεία η ερώτηση αυτή και δεν έχω παρά ένα λεπτό να απαντήσω. Θα εστιαστώ πρώτα απ' όλα στο ότι δεν έχουμε χάσει τη μάχη. Ε, σήμερα σε πολλές τεχνολογίες είμαστε ε, ηγέτες. Ε, ειδικότερα στις πράσινες τεχνολογίες μπορώ να σας διασφαλίσω είναι ήδη και θα συνεχίσει να είναι η πρώτη τεχνολογικά ήπειρος στον κόσμο. Είμαι πεπισμένος. Δεδομένου αυτό τώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε εξαρτώμεθα από κάποιες τεχνολογίες, αλλά οι προσπάθειες που έχουν γίνει και προηγουμένως μιλήσατε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμενας, οι προσπάθειες που έχουν γίνει από το Κοινοβούλιο σε αυτό τον κλάδο και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κρασνοτεύσκη για τις προσπάθειες που έχει κάνει ο συζητητής για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμενος. Είναι εξαιρετικά σημαντικές αυτές οι προσπάθειες που παρέχουν ε, τα μέσα ε, και θα σας περιγράψω τα μέσα που θα έχουμε για να αναπτύξουμε διτέ τεχνολογίες διπλής χρήση στο μέλλον. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Επόμενος ομιλητή Ντανίκα, εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιο επιτροπέ τις γραπτές απαντήσεις είπατε ότι θέλετε να είστε βέβαιος ε, και να διασφαλίσετε ότι η Ευρώπη θα υποστηρίξει τη βιομηχανική μας ε, ε, βάση για τη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία και ότι θα υπάρχουν εχέγγυα για τους πολίτες και για τις περιοχές που επηρεάζονται από την μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Δεδομένων των δυσκολιών που συναντάμε στις ε, περιοχές που πλήττονται περισσότερο από αυτή τη μετάβαση και σκεφτούμε αυτή τη στιγμή περισσότερο τις πλέον ενεργοβόρες βιομηχανίες. Ποια μέτρα θα προτείνετε συγκεκριμένα για να μειωθεί ο κίνδυνος ε, μετανάστευσης ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των βιομηχανιών μας. Με ποιο τρόπο θα συμμετέχετε εσείς σε αυτή τη δίκαιη μετάβαση ώστε να βρεθούν μηχανισμοί οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκή Βιομηχανία και που επίσης ε, θα διασφαλίσουν σε ίδιο επίπεδο την προστασία του επίπεδου ζωής ε, και του μέλλοντος των υπαλλήλων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Μπρέτον, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Νίτσα για την απάντησή σας. Είναι πολύ σημαντική. Προηγουμένως αναφέρθηκα σε μετάβαση ε, και αναφερόμαστε κυρίως εκεί σε, στη βιομηχανική μετάβαση. Πράγματι υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη πιο ευάλωτες από άλλες που μπορεί να πληγούν περισσότερο από άλλες ε, στη διάρκεια αυτή τη μετάβασης, κυρίως όσον αφορά τη βιομηχανική μετάβαση, τη βαριά βιομηχανία, Να σα δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Στην Ιταλία ε, που είχαμε ε, επί του θέματος, αλλά όχι μόνο. αφορούν η μετάβαση αυτή και περιοχές ή τομείς όπου υπάρχουν μετατροπές επαχθείς και εκεί υπάρχουν τα σχετικά ταμεία. Ε, τα σχετικά κονδύλια, τα οποία είναι εργαλεία πολύ εξειδικευμένα που μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξειδικευμένη βοήθεια σε, στα ενδιαφερόμενα κράτη, σε ενδιαφερόμενε περιοχές και να είστε βέβαιος ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσω προσωπικά. Γιατί όπως είπα προηγουμενω δεν μπορούμε να αφήνουμε οποιονδήποτε, ε, οποιονδήποτε ε, πίσω. Εάν είναι να έχουμε κανονε δεσμευτικου και αυτό είναι καλό που υπάρχουν, για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και κάποιες βιομηχανίες θέλουν να μεταφερθούν σε άλλα μέρη του πλανήτη όπου δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, τότε θα έχουμε αποτύχει. Οπότε υπολογίστε ότι βασιστείτε πάνω μου τα οικονομικά μέσα υπάρχουν. Θα το συζητήσουμε περισσότερο γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικότατο το θέμα και εγώ θα σταθώ σίγουρα στο πλευρό σας για να βοηθήσουμε αυτές τις περιοχές. Ξέρουμε ποιε είναι, είναι ορατές σήμερα καθαρά για να μπορέσουν να επωφεληθούν στο, κατά προτεραιότητα από αυτά τα οικολογικά κονδύλια για την οικολογική μετάβαση. Ευχαριστώ. Επερώτηση παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, πέραν αυτή τη δίκαιη μετάβαση, η ομάδα μας ε, έχει αγωνιστεί για το μηχανισμό προσαρμογής ε, άνθρακα. Διότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να ανταγωνιστεί την παγκόσμια βιομηχανία. Συναγωνίζεται βιομηχανίες που βρίσκονται σε χώρες όπου δεν έχει, δεν έχει θεσπιστεί κανένα μέτρο περιορισμού τη ρήπανση ή τέτοιο μέτρα δεν είναι προτεραιότητα και δεν φορολογείται η ρήπανση. Κατά συνέπεια, η δική μα βιομηχανία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Πιο συγκεκριμένα, κύριε υποψήφιε επίτροπε, πότε και πώς σκοπεύετε να υιοθετήσετε μέτρα για αυτόν τον μηχανισμό προσαρμογής στον άνθρακα. Ε, η ερώτηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Είμαι υπέρ αυτών των προσαρμογών. Διότι όπως είπατε πολύ σωστά, όχι μόνο προφυλάσσουν το περιβάλλον σε ολόκληρη μας την Ήπειρο, οπότε είναι κάτι καλό. Έχω εξετάσει σε βάθος τα ερωτήματα αυτά. Αλλά έχετε και δίκιο. Σήμερα, ε, και το είπα προηγουμένως ε, στην αναρκτήρια δήλωσή μου, πρέπει να μαχηθούμε. Ειδικότερα όταν έχουμε μπροστά μας αθέμητο ανταγωνισμό αυτό που είπατε είναι συγκεκριμένα παραδείγματα, τα γνωρίζουμε όλοι, όπου ο ανταγωνισμός πράγματι δεν είναι ισότιμος. Διότι οι χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν πρότυπα διαφορετικά από αυτά που επιθυμούμε εμείς για μας και για τους καταναλωτές μας. Ε, ένα από τα εργαλεία λοιπόν που θα είναι αυτός ο φόρο για τον άνθρακα που, στον οποίο αναφερθήκατε είναι ένα μέτρο το οποίο θα συζητηθεί. Εγώ θα το συζητήσω ανοιχτό μυαλά και ε, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη ομάδα Ρινιού, ε, η κυρία Χαράντσοβα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπρετόν, σας καλωσορίζουμε. Μας εξηγήσατε την καριέρα σας, το παρελθόν σας ε, και ε, είμαι σίγουρη ότι έχετε και την εμπειρία και τις ε, γνώσεις για να χειριστείτε καλά το χαρτοφυλάκιό σας. Αλλά θα ήθελα να γνωρίζω πώς θα χρησιμοποιήσετε την εμπειρία σας για να ολοκληρώσετε την κοινή αγορά. Η δέσμευσή σας ότι θα το κάνετε αυτό με τρόπο που να βοηθήσει όλα τα κρατημέλη, αυτό το ακούσαμε. Το τελευταίο κομμάτι της κοινή αγοράς είναι η πλήρης ε, η ελεύθερη μετακίνηση των υπηρεσιών. Ε, στην καριέρα σας ασχοληθήκατε με τέτοιες υπηρεσίες και ψηφιακές υπηρεσίες. Μήπως μπορείτε να πείτε στο Κοινοβούλιο πώς ακριβώς ε, προτίθεστε να επιτύχετε την ελεύθερη μετακίνηση υπηρεσιών και πώς θα επιτύχετε την πλήρη κοινή αγορά συμπεριλαμβανομένης και της κοινή αγοράς των υπηρεσιών. Ευχαριστώ πολύ. αγαπητή Ντίτα Τσαράντζοβα. Είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό θέμα και τα είπα λίγο και στην αρχή ότι οι υπηρεσίες είναι 70% του ΕΕΠ, πρόκειται για πολλές νέες θέσεις απασχόλησης, κάτι που είναι ζωτική σημασία. Ε, σήμερα τα όρια ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους παραδοσιακούς τομείς, γεωργία, βιομηχανία, αρχίζουν κάπως να μην είναι πια τόσο ξεκάθαρα. Οπότε, οφείλω να σας το πω από την αρχή θα είμαι σαφώς κατά κάθε νέου φραγμού. Είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα, το γνωρίζω. Μερικές φορές υπάρχουν, κάποιες χώρες τα θέλουν, δεν έπαιξαν πάντα το παιχνίδι όπως θα έπρεπε. Εγώ πάντως θα είμαι μαζί σας. Θα είμαι επίσης ξεκάθαρος ότι αν με ρωτάτε αν θα ξανανοίξω την οδηγία για τις υπηρεσίες, όχι. Αλλά θα φροντίσω να τεθεί σε εφαρμογή, γιατί υπάρχει και πρέπει να λειτουργεί, να γίνονται σεβαστοί κανόνες. Θα υπάρξει ίση μεταχείριση βεβαίως ανάμεσα σε όλες τις χώρες. Αυτό θα εφαρμόσω. Και έπειτα πέρα από όλα αυτά, εσείς αναφερθήκατε στα ψηφιακά, τα οποία αλλάζουν πολύ τα δεδομένα και είναι ένας μοχλός και αυτός που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να προσαρμόσουμε την οδηγία για τις υπηρεσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη κάνει πολλά. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευχαριστώ πολύ. Έχω ήδη δουλέψει για τα δεδομένα με την Επιτροπή μέχρι τώρα. Τώρα και πάλι θα πρέπει να τα ενισχύσουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να πάμε ακόμα πιο πέρα. Τώρα η πράξη για ε, τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι πολύ σημαντική. Έχει ήδη υπογραφεί από τις 28 χώρες. Θα φροντίσω για την εφαρμογή της, θα το επιβλέψω αυτό, γιατί βασίζομαι πολύ σε αυτή για να διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο τη ρευστότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών. Συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε στις ψηφιακές υπηρεσίες. Θα έχουμε την πράξη περί ψηφιακών υπηρεσιών και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τη θέλουμε αυτή την πράξη για να μην υπάρχει αυτή η κατάθμιση της αγοράς. Αυτή η ρήτρα περιορισμένης ευθύνη ήταν ε, καθοριστική σημασία για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών. Εσείς προτείνετε τέτοια πράξη να μην άρει, να μην αφαιρέσει αυτό το πολύ σημαντικό σκέλος ε, της οδηγίας περί ηλεκτρονικού εμπορίου. Απάντηση. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το διευκρινίσω. Ναι, δεν θα την πειράξουμε. Δεν θα την αμφισβητήσουμε. Όμως είδα ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες που βέβαια δεν προχώρησαν στο προηγούμενο κοινοβούλιο. Τα ξέρω αυτά. Εγώ έρχομαι εδώ με νέο πνεύμα. Θα κοιτάξω. Γιατί δεν προχώρησε. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν δεσμεύομαι, αλλά σίγουρα θα το κοιτάξω. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβη και να μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Τουσάν εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Καλημέρα κύριε Μπροτό. Αν αναλάβετε καθήκοντα θα αναλάβετε και ένα χαρτοφυλάκι, το οποίο θα καλύπτει τη βιομηχανική πολιτική, τον ψηφιακό τομέα, την άμυνα, το διάστημα και την εσωτερική αγορά ταυτόχρονα παραδεχτείτε ότι πρόκειται για μια τεράστια δύναμη, όπω και οι ανησυχίε μα είναι τεράστιε, διότι αυτέ οι επιχειρήσει που έχετε διευθύνει μέχρι πρόσφατα ε, δραστηριοποιούνται στο σύνολο των κλάδων που μόλι ανέφερα. Και το βλέπουμε πώ επικαλύπτονται όλοι αυτοί οι κλάδοι. Η αλήθεια είναι ότι η υποψηφιότητά σας αποτελεί ένα μείγμα που δημιουργεί σύγχυση σε εποχέ που χρειαζόμαστε καθαρότητα ε, ε, προ υπερασπιση του κοινού συμφέροντο. Όταν ήσασταν υπουργό οικονομία στη Γαλλία, ε, είχατε ε, απορρίψει φακέλου που θα μπορούσαν να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο και εδώ. Αναλαμβάνετε δεσμεύσει ότι θα υπερασπίζετε το γενικό συμφέρον και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα. Γενικό συμφέρον είναι μια Ευρώπη που μάχεται κατά τη κλιματική αλλαγή. Οι ευθύνε σα ε, ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό το ψηφιακό κλάδο. Αλλά ε, ω πολιτικό απαντήσατε μόνο σε αυτό, για αυτόν τον κλάδο. Τι θα κάνετε για τη σύγκρουση συμφερόντων ε, και για να ε, προωθήστε την Ευρώπη στην ε, υπεράσπιση των οικολογικών της συμφερόντων. Ευχαριστώ που μου θέσετε αυτή την ερώτηση. Είναι κάτι που με έχει απασχολήσει πολύ. Ε, το έθεσα και στην αρχική μου ομιλία και έχετε δίκιο που με ρωτάτε κάτι τέτοιο. Γιατί πράγματι αυτή η έννοια βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης μου. Ανέκαθεν ήταν έτσι. Κάθε φορά που αναλάμβανα καθήκοντα, τα αναλάμβανα 100%. Γι' αυτό ήρθα μπροστά σα, χωρί κανέναν δεσμό πλέον, οποιοδήποτε είδο με την επιχείρηση που δίθυνα. Κανέναν δεσμό, όπω είπα. Φυσικά ε, πρέπει να δούμε και ποιε είναι οι προθέσει. Ε, ε, ο κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει προβλέψει στο άρθρα 2 και 6 και 4 του κώδικα υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί ώστε άνθρωποι όπως εγώ, όπως άλλοι, σαν εσά που μπορεί να προέρχονται από από, την, ε, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από δικηγορικά γραφεία να μπορούν μια μέρα να βρεθούν σε αυτή τη θέση. Αλλά πρέπει να το πούμε σαφώ φυσικά ε, στη διακυβέρνηση. Και το λέω, θα είμαι ε, ρηξικέλευθος, θα εφαρμόζω κατά γράμμα αυτή την αρχή. Σίγουρα υπήρξαν κάποιες επαφές μεταξύ των επιχειρήσεων που διεύθυνα και της Κομισιόν. μα αυτό είναι φυσιολογικό. και θα υπάρχουν ε, τέτοιες. Ε, ξέρετε, και, ακόμη και διαγωνισμοί, όλα αυτά γίνονται με διαφάνεια. αυτό ο οίκο, εδώ το κοινοβούλιο και η θέση μου αύριο είναι ε, μέρη όπου τα πάντα καταγράφονται, όλα τα ραντεβού. Και το γνωρίζετε αυτό και μπορεί, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να βλέπετε τις πληροφορίες. Οπότε, εάν κάποια στιγμή κάποιο ζήτημα απαιτεί την παρουσία ε, και τη συμμετοχή του ε, Επιτρόπου. Σύμφωνα με αυτά τα δύο άρθρα, η Πρόεδρος ε, επικαλείται αυτά τα δύο άρθρα και έτσι καθορίζεται ποιος Επιτρόπος θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα όταν απαιτείται παρουσία του Επιτρόπου. Θα είναι απλά τα πράγματα, σαφή και ακριβή. Συγγνώμη για το δεύτερο κομμάτι. Ευχαριστούμε. Συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Τουσά. Να ευχαριστώ για την απάντησή σας. Ωστόσο, έχω κάποιες αμφιβολίες γιατί αυτό δεν το είδατε το σα σας έδειξα το σχήμα. Υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των δραστηριοτήτων σας. Όταν λοιπόν δεσμεύεστε να μην λαμβάνετε αποφάσεις σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες, θέλω να με εξηγήσετε καλύτερα πώς ε, σκοπεύετε να το κάνετε αυτό. Και μετά ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση για την βιομηχανική πολιτική που θα εφαρμοστεί για να καταπολεμηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη και η έλλειψη των πόρων. Θα μπορούσατε να μου απαντήσετε λοιπόν συγκεκριμένα. Θα μου κάνατε μεγάλη χαρή. Ευχαριστώ. Πρώτον, πρώτη ερώτηση, αγαπητή κυρία. Ε, δεν ε, θα ε, επικαλύπτω ένα τομέα με τον άλλο. Δεν θα ξεφύγω από τους τομείς που θα έχω αναλάβει στο ψηφιακό κόσμο, στα ηλεκτρονικά, στις τηλεπικοινωνίες. Πιστέψτε με, πάντα δρούσα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και ούτως θα πράττω και τώρα. Σε περίπτωση που χρειαστεί να πάει ο Επίτροπος ε, για συμβάσεις, για επιχορηγήσεις. Οι συμβάσει μεταξύ της Άτος ε, και της Κομισιόν ε, το 2018 αναρχόταν σε 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 0,01% του κονδυλίου που παρέχεται για τις επιχειρήσεις. Οπότε θα λειτουργώ με αυστηρότητα και μόνο για τα θέματα που ανέφερα και σίγουρα όχι για το σύνολο του χαρτοφυλακίου. Κατά τα άλλα, η πράσινη πολιτική βρίσκεται στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μου. Θα ε, ε, εστιαστούμε στι ε, τεχνολογικέ μετάβαση και θα το ξανασυζητήσουμε αργότερα στην ακρόαση. Γιατί, όπω είπα, είναι ένα θέμα όπου η Ευρώπη πρέπει, είναι υποχρεωμένη και θα νικήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μελά. Έχει τώρα το λόγο εκ μέρου τη ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι καταλαβαίνετε πως η αποστολή σας θα διεξαχθεί μέσα σε ένα προβληματικό πλαίσιο, μια εσωτερική αγορά που έχει φτάσει στα ωριά τη, με κανόνες ανταγωνισμού που καθόλου παρά ισότιμοι είναι, με ρυθμίσεις όσον αφορά τις δημόσιες αγορές κλπ. Μια Ευρώπη που έχει γεράσει, που έχει χάσει τη νιώτη της και το σφρίγο της και βρίσκεται σε κατάσταση εκτός ελέγχου. Όσο λοιπόν επίτροπος για το χαρτοφυλάκιό σας, σίγουρα ε, θα βρεθείτε αντιμέτωπος με όλα αυτά και ίσως θα έπρεπε η αποστολή σας να είχε δοθεί σε διαφορετικά άτομα, να είχε μοιραστεί κάπως για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τα νομοθετικά κείμενα. Τώρα, επίσης, θα πρέπει να είσαστε αποτελεσματικό και σε πράγματα όπως είναι το Ταμείο της Άμυνας, όπου έχει μείνει πάρα πολύ πίσω η Ευρώπη, όπως επίσης και για την τεχνητή νοημοσύνη, το 5G, όπου βρισκόμαστε πολύ πιο πίσω από Κινέζους και άλλους. Συνεπώς, κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, πώς εσείς θα οργανωθείτε, πώς θα χρηματοδοτήσετε, πώς θα δικαιολογήσετε απέναντι στους πολίτες τους κύριους αυτούς άξονες της εντολής σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευρωβουλευτή. Η ερώτησή σας πράγματι βρίσκεται στην καρδιά του χαρτοφυλακίου μου. Γιατί βλέπετε, ας σταθούμε λίγο, ας σταθούμε. Τι μήνυμα στέλνουμε στον υπόλοιπο κόσμο. Αν επιβεβαιώσετε την ε, εντολή μου, θα στείλουμε το μήνυμα ότι στην Ευρώπη Έχουμε καταλάβει ότι για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μετάβασης και των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να υπάρχει μία ενιαία εντολή, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, στα θέματα που τροποποιούν τη δραστηριότητά μας, τη βιομηχανία μας, τη ζωή μας. Δηλαδή ψηφιακή τροποποίηση και οικολογική φιλοδοξία. Είναι δύο άξονες οι οποίοι θα διαρθρώσουν τις τεχνολογικές, βιομηχανικές και επιστημονικές εξελίξεις μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Συνεπώς, εδώ στις Βρυξέλλες είναι που θα έχουμε αποφασίσει να έχουμε μία πράξη εντολή, η οποία θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Αυτό θα είναι το μήνυμα που θα στείλουμε. Όσον αφορά εμένα, ξέρω ότι το χαρτοφυλάκιό μου είναι ιδιαίτερα ευρύ Πριν αναφερθήκατε στο γεγονός ότι ήμουνα υπουργό Οικονομίας, Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Τουρισμού σε μια κυβέρνηση που ήταν ε, ακόμα ευρύτερη. Δεν είναι ότι συγκρίνω, αλλά απλώς το λέω γιατί πρέπει κανείς να είναι σε θέση να διαχειριστεί το σύνολο των προκλήσεων και εγώ θα χρησιμοποιήσω όλη μου την ενέργεια προς αυτό το σκοπό. Ευχαριστούμε. Συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Ε, σημείωσα ότι όσο και έλαφρος εσείς μας παρουσιαστήκατε ε, για τη σύγχρονη οικονομία που γνωρίζει τις δυσκολίες, τις σημερινές, τις ευρωπαϊκές, τις εθνικές, ε, παγκόσμιες κτλ. Όμως νομίζω ότι εδώ κρύβεστε πίσω από μία γενικόλογη συνένεση και τα μπερδεύετε όλα και όλες τις ταυτότητες. Οπότε ακόμα και αν τεχνολογικά οι γνώσεις σας είναι ενδιαφέρουσες και φαίνεται αυτό από τη σταδιοδρομία σας, κατά τη γνώμη μας αυτό δεν φτάνει. Αν δεν υπάρχει περισσότερη ουσία γύρω από τα λόγια, τότε όλα αυτά είναι περίτα. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε έναν πραγματικά καλό λόγο για τον οποίο η ομάδα μας να μην απορρίψει την υποψηφιότητά σας. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Κοιτάστε, είπατε ότι είμαι ρηξικέλαθρος, ναι. Κοιτάξτε, το θέμα της διακυβέρνησης και της διαχείρισης είναι κάτι που με παθιάζει. Σε όλη μου τη σταδιοδρομία το έκανα. Είναι αναγκαίο να υπάρχει μια αυτονομία, μια ανεξαρτησία η οποία να προστατεύει την ε, εντολή και τα καθήκοντα. Και εδώ βρίσκομαι μπροστά σας γιατί στην προηγούμενη σταδιοδρομία μου αυτό το κατάφερα. Αυτό ήταν ο στόχος μου. Επίσης έχω διδάξει και διακυβέρνηση σε ένα Αμερικανικό Πανεπιστήμιο γιατί μου αρέσει το θέμα αυτό. Το βάζω και στην ε, πράξη. Το κάνω πράξη, το εφαρμόζω. Διάκριση εξουσιών, βεβαίως. Από εκεί και πέρα, εσείς πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να γίνει. Ο καθένας στο δικό του ρόλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους ε, της ομάδας ECR, Adam Μπίλαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία από τις αποτυχίες της Επιτροπής Juncker ήταν η αδυναμία να προχωρήσει στον τομέα των παραδοσιακών υπηρεσιών. Ε, πριν από ε, κάποιες εβδομάδες ε, και αυτό που ακούσαμε δεν μας προσέφερε πολλές ελπίδες. Η τεχνολογική κυριαρχία και η νέα κούρσα στο διάστημα. Αυτά είναι νέες ιδέες, αλλά εμείς έχουμε έναν παραδοσιακό τομέα υπηρεσιών και εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες και πάρα πολλοί πολιτικοί που υπογραμμίζουν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Όμως όσον αφορά στην εναρμόνιση της αγοράς, όλοι αυτοί κρύβονται πίσω από προστατευτικούς αγωνισμούς και φοβούνται τον θεμητό ανταγωνισμό. Με βάση την προηγούμενη απάντησή σας, δεν αρκεί μόνο να εμποδίσουμε να εμφανιστούν εμπόδια, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και εμπόδια που ήδη υπάρχουν τώρα. Ε, θέλω να πιστεύω ότι εσείς ε, θα βοηθήσετε στο να ε, διαχυθούν οι υπηρεσίες ε, στο λιανικό εμπόριο, στο χοντρικό εμπόριο, σε πάρα πολλούς τομείς, γιατί οι επιχειρηματίες και οι πολίτες δεν μπορούν πια να ακούνε άλλες δικαιολογίες. Έχει φτάσει για μας εποχή να ανασκουμποθούμε και γι' αυτό χρειαζόμαστε την δική σας τη δέσμευση και την υποστήριξη. Ευχαριστώ. Έχει συζητηθεί και θα ξανασυζητηθεί πολύ το ζήτημα αυτό. Βρίσκεται στο επίκεντρο του χαρτοφυλακίου φυσικά που θα αναλάβω εγώ αν με επιβεβαιώσετε σε αυτή την αποστολή, σε αυτό το λειτουργήμα. Όπως είπα, πρέπει να εργαστούμε με αυτά που έχουμε. Συμμερίζομαι την ανάλυση σας και συμφωνώ. Έχω ήδη πει ότι θα μαχηθώ κατά των περιφερειακών προστατευτισμών. Βλέπω κι εγώ, όπως και εσείς, ότι υπάρχουν φραγμοί. Είναι σαφές. Θέλω να είμαι ρεαλιστή και όχι δογματικό. Και επίση θέλω να εστιαστώ εκεί όπου μπορούν να σημειωθούν πρόοδοι το συντομότερο δυνατόν το ταχύτερο. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσω να σταθώ στο πλάι σας. Ναι, το, αναλαμβάνω τη δέσμευση με μεγάλη μου χαρά μπροστά σας. Θα είναι ένα τεράστιο διακύβευμα ε, για το οποίο θα δεσμευτώ. Πέραν αυτού τώρα υπάρχει και το θέμα της ε, ελευθερίας του επιχειρήν σε σχέση με τον προστατευτισμό ε, και την προστασία, όλα τα προβλήματα απάτης και εγώ θα πάω να ψάξω να δω τι συμβαίνει, να υπάρξουν κάποιες κυρώσει. Και υπολογίζω, ε, σκοπεύω να χρησιμοποιήσω αυτή την εξουσία που θα μου ανατεθεί ε, και θα ήθελα να το ξέρετε εδώ, για την εφαρμογή των κανόνων. Έχει έρθει η ώρα για να γίνει κάτι τέτοιο. Προηγουμένως ε, αναφερθήκατε στις ψηφιακές υπηρεσίε. και θέλω να πω ότι βλέπω κάτι εντελώ καινούριο, εξαιρετικό. Επιτέλους Αντί να πηγαίνουν από Ανατολά προ Δυσμά, πάνε τώρα από Δυσμά προ Ανατολέ. Προ Ανατολέ και ειδικότερα στι υπηρεσίε ε, υψηλοτερη προσθέμενη αξία ε, του ψηφιακού κόσμου. Η Πολωνία έχει αναπτύξει πολύ την ψηφιακή ασφάλεια, το ίδιο και η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και τώρα έχουμε αμφίδρομη πλέον ροή. Είναι καλό σημάδι και το ενθαρρύνω. Και θα το ενθαρρύνω επίση. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, συμπληρωματική ερώτηση κύριε Μπιέλαν. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή έχετε εμπειρία, ε, ήσασταν επικεφαλής ψηφιακής επιχείρησης. Κατά την άποψή ποιοι είναι οι πιο δύσκολοι κανονισμοί οι οποίοι ε, καθυστερούν την εξέλιξη μιας εταιρεία όπως της Άτος και της αλυσίδας παραγωγής. Ε, θέλω να ρωτήσω κατά πόσον έχετε κάποιες επιθυμίες που έχετε κατά νου για να αλλάξετε την αγορά. Η κυρία Γκουλάρ είπε ότι ε, θέλει κατά τη διάρκεια, των νομοθετικών κατά τη διάρκεια της νομοθετικής της ε, θητείας να προσπαθήσει να βρει λύση σε αυτά τα προβλήματα που θα ξανατεθούν. Εσείς τι πιστεύετε από αυτού. Επιτρέψτε μου να απαντήσω γενικά στην ερώτησή σας και να σας πω μόνο ότι ε, διαπίστωσα σε διάφορους κλάδους και θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε στο πλαίσιο της περιπολιτικής περί ανταγωνισμού και θα πρέπει να την αναθεωρήσουμε δεδομένου τη ψηφιακή τεχνολογία. Βλέπουμε κάποιου μεγάλου ομίλου στην Ευρώπη. Αυτό ε, από τον οποίο μόλι έφυγα εγώ είναι ένα παράδειγμα. Και υπάρχουν και τα τεράστια κονδύλια τη σχετική γενική διεύθυνση. Οι κανόνε είναι υπαρκτοί. Υπάρχει και ο ελεύθερο ανταγωνισμό. Το πρόβλημα όπου προσκρούμε είναι ότι δεν είναι τόσο για του μεγάλου ομίλου, άρα περισσότερο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και το βασικό πράγμα που με απασχολεί είναι οι μικρομεσαίε. Επιχειρήσει αυτέ υποφέρουν, αυτέ δεν έχουν τα μέσα. Οι μεγάλε επιχειρήσει έχουν τα μέσα. Αλλά οι μικρομεσαίε επιχειρήσει έχουν ελάχιστα πόρου. Οπότε ε, θα εστιαστώ στο πώ θα τι ε, βοηθήσω. Θα έχω κάποιον εντεταλμένο που θα πηγαίνει επί τόπου να βλέπει τι γίνεται για να ε, μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε τα σημεία συμφόρηση. Αυτό. Θέλουμε να απελευθερώσουμε την εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Εκ, ε, εκ, εκ μέρους της Γκουε, ο κύριος Μπόμπα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπρετόν, ω Γάλλο βουλευτή πρέπει να σα πω ότι αισθάνομαι πολύ αβόλα, διότι το χαρτοφυλάκιο στο οποίο αναφερόμαστε τώρα είναι σημαντικό και λόγω της συνοχής ε, αλλά και γιατί σήμερα δεν μπορείτε να μου πείτε ότι οι παρελθούσε δραστηριότητε σα δεν θα ε, επηρεάσουν τι μελλοντικέ σα αποφάσει. Κοιτάτε, λέτε ότι δεν θα αναμειχθείτε σε φακέλου που θα αφορούν την επιχείρηση ΑΤΟ. Γιατί μιλάμε. υποστήριξη προ τη βιομηχανία. Η Άτος πήρε το 2018 πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το, η ψηφιακή τεχνολογία θα έχετε να ασχοληθείτε με την ανάπτυξη των υπερυπολογιστών που θα έχουν ένα κατασκευαστή στην Ευρώπη την παλιά σα επιχείρηση, την εσωτερική αγορά θα πρέπει να ε, καταπολεμήσετε το παράνομο εμπόριο οπουδήποτε, αφού έχετε δημιουργήσει ένα σύστημα χνηλάτιση για τη Φίλιπ Μόρι. Για την άμυνα, όταν η Άτο ε, ε, παίζει σημαντικό ρόλο στη στρατηγικό εξοπλισμό. Στην άμυνα, ίδιο, ενώ συμμετέχει στο, και στο διάστημα συμμετέχει η Άτο στο Κοπέρνικου. Αυτή η σχέση με την παλιά επιχείρηση που λέτε, αν πάψουν να υπάρχουν, δεν θα έχετε χαρτοφυλάκιο, δεν θα έχετε καμία επιρροή. Οπότε η ερώτησή μου είναι η εξή. Σήμερα ζητάτε η θέση του Γάλλου Επιτρόπου να είναι μια θέση πλαστή. Ε, παρακαλούμε απαντήστε. Ευχαριστώ κύριε Μπομπά. Θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Τρία στοιχεία. Πρώτον, ουδέποτε είπα, παίξατε με τα λόγια, δεν είπα, είπα ότι σαφώς αφού υπάρχει κανονισμός ε, τα άρθρα 2, 6 και 4 ε, του κανονισμού της Κομισιόν. Αν υπάρχουν οποιασδήποτε σχέσεις μπορείτε να με απορρίψετε. Ας μην παίζουμε ε, με τα λόγια. 100 ε, εκατομμύρια κύριε Μπομπά. Μιλάτε για την HPC και Codify 100 εκατομμύρια. Όχι, κάνετε λάθος. 135 το 2018. Και γιατί 135. Διότι 37 εκατομμύρια ευρώ κλασικές παροχές μεταξύ ε, Κομισιόν και Άτος 90 ε, με όλους τους φορείς αεροκοντρόλ, διαγωνισμοί που έγιναν φυσικά δημόσια και μετά 16 εκατομμύρια επιχορηγήσεις, όχι 100 για 102 προγράμματα, δηλαδή 500.000 ευρώ ένα πρόγραμμα μόνο που εκχωρήθηκαν μόνο μετά αφού τηρήθηκαν οι κανόνες ανταγωνισμού και αγοράς ε, για τις υπηρεσίες. Η επιχείρηση αυτή, η αεροσπασία που αναφέρεται, είναι επιχείρηση. Αυτή έκανε τα ε, ε, σύναψη τη συμβάση, όχι η Κομισιόν και μετά αν υπάρξει κάποιο διαγωνισμό και αφορά την ΝΑΤΟΣ, δεν θα ενημερωθώ. Είναι πολύ απλό. Και τέλος, αναφέρεστε στην καπνοβιομηχανία, εγώ δεν την γνωρίζω καθόλου. Αναφέρεστε στο Codify που είναι ένα σύστημα εχνηλάτησης το οποίο αγόρασε η Άτος όταν ε, ξέρω τη Siemens μια λυσίδα, τη World Line, που δεν είναι σήμερα άτο, είναι απλά μια θηγατρική, δεν υπάρχει ούτε Ουδέποτε συνάντησα εγώ ανθρώπου από την καπνοβιομηχανία, ούτε από κοντά ούτε από μακριά. Οπότε η αυτονομία μου, σα το εγγυώμαι, θα είναι απόλυτη και θα είμαι επίτροπο για, όλα τα, για όλε τι πτυχέ του χαρτοφυλακίου. Παρακαλώ, συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Μπομπά, κύριε Μπρετό, Αναφέρετε το κώδικα διοντολογία των επιτρόπων. Λένε ότι οι επίτροποι σε οποιαδήποτε κατάσταση όπου υπάρχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων ε, θα πρέπει να εξετάζεται ως τέτοια αυτή η περίπτωση. Εμείς ε, ως Ευρωπαίοι πολίτες πώς μπορούμε να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος όταν φύγατε από μια επιχείρηση και όπου πουλήσατε τις μετοχές σας για 40 εκατομμύρια ευρώ όταν λέτε ότι δεν θα ασχοληθείτε με πτυχές που θα αφορούν αυτή την επιχείρηση αυτό αφορά και τους ανταγωνιστές τους ε, ε, πιθανούς εταίρους αυτής της επιχείρησης ε, προγράμματα που ενδεχομένως να έχετε από κοινού, όπως βλέπετε, είναι απαράδεκτο. Πριν από ένα μήνα απορρίψαμε την κυρία Γκουλάρ. Κύριε Μπρετόν, για ποιο λόγο, και η ερώτηση απευθύνεται σε εσά και στους συναδέλφους μου όμως, για ποιο λόγο θεωρείτε σήμερα ότι αυτό που απορρίψαμε πριν από ένα μήνα πρέπει να το δεχτούμε σήμερα. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι θα πρέπει εσάς να σας δούμε πιο ευνοϊκά. traitement de faveur. Κύριε Μπομπά, καμία ευνοϊκή μεταχείριση, μηδέν, μηδέν ευνοϊκή μεταχείριση. Κάντε ό,τι θέλετε. Εσείς θα με επιβεβαιώσετε, εσείς θα, με νομιμοποιήσετε. Κάντε αυτό που επιθυμείτε και εγώ θα το σεβαστώ. Σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά εγώ δεν περίμενα να αποφασίσετε εσείς. Έδρασα προκαταβολικά. Ήθελα να πω σε όλους τους ε, συμπολίτες μας και όχι μόνο τους Γάλλους, κύριε Μπομπά. Είπα, θέλω να έρθω ενώπιον σας, ανεξαρτήτως της απόφασης που θα λάβετε εσείς, ε, έχοντα ε, εγκαταλείψει όλα μου τα λειτουργήματα, όλε μου τι θέσει και όλε μου τι μετοχέ στην αγορά. Και εσεί μετά θα αποφασίσετε. Εγώ ανέλαβα τι ευθύνε μου. Είμαι απολύτω ανεξάρτητο. Αλλά μην το επαναλαμβάνετε. Δεν πρόκειται να ξαναμεταφερθώ στον κλάδο αυτό. Ε, θα ε, συμπεριφερθώ μόνο βάσει του κώδικα, κύριε Μπομπά, διότι θα υπάρχουν συμβάσεις, πράγματι και οικονομικές σχέσεις που θα έρθουν σε μένα, αλλά που δεν θα τις γνωρίζω, δεν θα πρέπει να τις γνωρίζω και θα το κάνω με απόλυτη ανεξαρτησία, εξυπηρετώντας τα γενικά ευρωπαϊκά συμφέροντα. Um, uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ντεσούτερ Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ο γύρος των ερωτήσεων από πολιτικές ομάδες, από εκπροσώπους πολιτικών ομάδων και τώρα θα συνεχίσουμε με μεμονωμένους ε, ευρωβουλευτές. Ο πρώτος είναι ο κύριος Σουβάπ από την ΙΜΚΟ. Παρακαλώ κύριε Σουβάπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, Άκουσα πόσο ξεκάθαρος ήσασταν όσον αφορά το γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Και θέλω να σας πω ότι θέλω λιγάκι να σας προκαλέσω, γιατί αν θεωρείτε ότι η κοινή αγορά είναι μια μεγάλη αγορά που επιτρέπει σύγκληση και ανάπτυξη, θα πρέπει όμως να πούμε και ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας τέτοιος ανταγωνισμός που να αφορά όλα τα κράτη και όλες τις επιχειρήσεις. Επειδή λοιπόν το έχετε πει και έχει υποθεί επανειλημμένα, να σας πω κάτι. Το ΕΛΚ είναι υπερήφανο για κάθε επιτυχημένη επιχείρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε με την νομοθεσία κοινή αγορά να βοηθήσουμε επιχειρήσει ακόμα περισσότερε να έχουν επιτυχία. Ήρθατε όμω εδώ στι Βρυξέλλε για κάποια συγκεκριμένη δουλειά και γι' αυτό θέλω να σα πω μία μικρή ιστορία, να σα δείξω πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Εδώ στι Βρυξέλλε φιλοξενούσα ε, προέδρου ε, πρωθυπουργού ε, και αυτοί λοιπόν όταν ήθελαν να κάνουν συζητήσει και συναντήσει έπρεπε να συμπληρώσουν το έντυπο Α1. Αυτό δυσκολεύει τη ζωή μα στην Ευρώπη και και γι' αυτό ρωτάω, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε αυτό το έντυπο να καταργηθεί επιτέλους, να ανήκει στο παρελθόν. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Πολλές ερωτήσεις, κύριε Ευρωβουλευτά. Αλλά εντάξει. Ξέρω ότι είναι θέματα που σας απασχολούν πολύ και σας ενδιαφέρουν. Ανταγωνισμός, ουσιαστικά, έτσι. Η ερώτησή σας αυτό είναι. ανταγωνισμός. Πώς θα έχουμε σωστό, υγιή, λογικό ανταγωνισμό στην Ευρώπη και, μια που αναφέρεστε στην Φόρμουλα 1, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να υποφελουθούν όπως και οι άλλοι. Τώρα, επειδή είναι ευρεία η ερώτησή σας, εγώ θα επικεντρωθώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, ειλικρινά πιστεύω ότι οι κανόνες ανταγωνισμού δεν είναι ακόμα αρκετά προσαρμοσμένη στη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και ναι, το έντυπο αυτό που λέτε αποτελεί μία περίπτωση, το έντυπο 1, και μιλάω, όχι μόνο από εμπειρία, όταν ήμουν εγώ πιο νέος έφτιαξα μια μικρομεσαία επιχείρηση και όταν κανείς είναι μόνος του είναι πιο εύκολο. Όταν όμως έπρεπε να προσλάβω τον πρώτο μου υπάλληλο, τότε ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί η ζωή του εξαρτιάται από εσά που έχετε την επιχείρηση. Υπάρχει η υπερβολική τεχνοκρατία. Από την άλλη μεριά προσπαθείτε να μεγαλώσετε όταν είσαστε μικρομεσαία επιχείρηση. Προσπαθείτε να συμμετέχετε στις δημόσιες αγορές, κάτι το οποίο δεν γίνεται αρκετά σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκο να έχει πρόσβαση μια μικρομεσαία ε, στις δημόσιες προσφορές. Οπότε, όσον με αφορά, όλες οι πτυχές που μπορούν να βοηθήσουν να υπάρξει διέξοδος όλα αυτά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την ευρία έννοια, θα το κάνω. Να είσαστε σίγουροι. Γιατί δεν θέλω να υπάρχει τροχοπέδι στον ανταγωνισμό. Και είπαμε ότι το 99% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Η συμπληρωματική ερώτηση του κύριου Σφάβα. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Αυτό όμω σημαίνει ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να επιτρέπουμε τον ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να δημιουργήσουμε θεμητέ και δίκαιε συνθήκε ανταγωνισμού για όλους. Και αυτό είναι δύσκολο για τα επόμενα χρόνια. Βλέπουμε ότι ο πλούτος κατανέμεται διαφορετικά στο βορρά, στο νότο, στην Ανατολή, στη Δύση. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε έτσι ώστε να προσφέρουμε προοπτική για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, να νιώθουν ότι αξίζει η δουλειά τους διότι έχουν την προοπτική να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Εδώ με ρωτάτε το βασικό. Είμαστε μία Ήπειρος. Ήπειρος η οποία τις διαφορές μας, την ιστορία μας και τις πιο πρόσφατες ιστορίες μας τις συγκέρασε. Υπάρχουν διαφορές ακόμα Ανατολή, Δύση, Βορράς, Νότος. Ακριβώς επειδή τα βλέπω όλα αυτά, μια που μου ζητήθηκε να έρθω εδώ, μου το πρότεινε η κυρία Φοντερ Λάιεν, το δέχτηκα. Γιατί όντως η τροχοπέδρα είναι μεγάλη. Το καλό είναι όμως είναι ότι μπορούμε, ξέρουμε πώς θα τα καταφέρουμε και οι δυνατότητες που έχουμε να απελευθερώσουμε όλο αυτό το δυναμισμό που υπάρχει είναι τεράστιες. Τις τελευταίες ε, μέρες συναντήθηκα με καμιά πενταριά από και όλοι σας βοηθήσατε. Κατάλαβα ποιες είναι οι ανησυχίες σας, κατάλαβα ποιοι είναι οι προβληματισμοί σας. Και εσείς είσαστε οι εκπρόσωποι του κόσμου, οπότε καταλαβαίνω. Και κάθε φορά που κάτι μπορεί να γίνει, κάποιος από εσά έχει το κλειδί για να ξεκλειδώσουμε κάτι, να μου το δίνει παρακαλώ. Ακριβώς για να ξεκλειδώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν τροχοπέδι και εμποδίζουν την πρόοδο στην Ευρώπη. Η κυρία Σαλντεμόζ είναι επόμενη από τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπρετόν. Το γραπτό ερωτηματολόγιο που σας δόθηκε ε, αναφέρεστε στην κυρία Φοντελάιν που αναφέρει ότι εγώ πιστεύω σε μια Ευρώπη η οποία μπορεί να συμφιλειώσει το κοινωνικό στοιχείο με την κοινωνική αγορά. Μια Ευρώπη όπου όλοι θα μπορούν να επιτύχουν πολλά πράγματα. Και εσείς λέτε ότι θα δουλέψετε για μια κοινή αγορά που θα είναι ε, στην υπηρεσία των πολιτών. Και σήμερα είπατε ότι δεσμεύεστε να μην αφήσετε κανέναν σε μειονεκτική ε, θέση. Αυτά μοιάζουν λόγια σοσιαλδημοκρατών. Αλλά βλέποντας τα προγράμματά σας δεν βλέπω τίποτα το συγκεκριμένο προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπω προγράμματα για τις επιχειρήσεις, αλλά δεν βλέπω να προτείνετε τίποτα για το κοινωνικό στοιχείο. Μήπως μπορείτε να μας πείτε λιγάκι πώς θα δουλέψετε για μια κοινωνική Ευρώπη, μια Ευρώπη που θα δουλεύει προς όφελος όλων και δεν θα παραμελεί κανέναν. Ο κύριος Μπρετόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαλντεμόζε. Από τις συζητήσεις μας Ξέρω ότι σας απασχολεί αυτό το θέμα, το υπενθυμίσατε, αλλά και εμένα. Γιατί το είδατε. Το υπενθύμισα πριν η τρίτη πρόκληση είναι ο δικός μου ο άξονας. Τρίτη πρόκληση το ονόμασε η εκλεγμένη πρόεδρος. Όντως είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε τους πάντες. Θα συνεργαστούμε. Αν μη τι άλλο τίτλος του χαρτοφυλακίου που ελπίζω να αναλάβω, έχει εξελιχθεί. Το είχε ο κύριο Σμιτ πριν. Οπότε έχουμε μιλήσει αρκετά. Θα συνεργαστούμε. Ο κύριος Σμιτ θα είναι ο κύριος μου συνομιλητής. Εγώ τώρα τι μπορώ να προσφέρω. Πρώτα απ' όλα ε, κονδύλια, κόμβους που σκοπεύω να τους αναπτύξω περισσότερο προβλέπονται ήδη. Θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και όλους όσοι θέλουν να φροντίσουν να υπάρχει δουλειά πιο κοντά εκεί που βρίσκονται. Γι' αυτό θα φροντίσουμε να δημιουργηθούν αυτοί οι κόμβοι με την κατάλληλη χρηματοδότηση βέβαια. Θέλω όμως να πάω και ακόμα πιο μακριά. Γιατί αυτή η κοινωνική διάσταση έχει να κάνει και με νέα, νέες δουλειές. Ε, για παράδειγμα με τη μορφή πλατφόρμων. Ξέρετε για τις πλατφόρμες όπου βλέπουμε τα πάντα. Δεν ε, προστατεύουμε όπως θα έπρεπε ε, και δεν δίνουμε τις εγγύσεις που θα έπρεπε. Οπότε και εγώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της θα φροντίσουμε ώστε να τηρούνται κανόνες ώστε και αυτοί που εργάζονται στις πλατφόρμες αυτές, που είναι κάπου 10% ε, των Ευρωπαίων εργαζομένων που τη μια την άλλη μέρα πέρασαν από τέτοιες πλατφόρμες. Γι' αυτό λοιπόν θα φροντίσουμε να υπάρχουν πληροφορίες, ευαισθητοποίηση ότι χρειάζεται και κατάλληλη χρηματοδότηση. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε αυτέ τι νέε θέσει απασχόληση που είναι και διαφορετικών μορφών πολλέ φορέ. Για συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Σάλντε Μόγερ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να συνεχίσω διότι όταν εργαζόμαστε με την εσωτερική αγορά προσπαθούμε να άρουμε τα σπεριτούς φραγμούς και ε, το είπατε κι εσείς, αυτή ήταν μια ιδέα που είχατε για ε, να κάνουμε κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά πώς θα γίνει αυτό ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων. Γιατί πολλές, ε, πολλά από τα εμπόδια που έχουμε στην κοινή αγορά έχουν ως στόχο να προστατεύουν τους καταναλωτές. Λοιπόν, ε, εσείς λέτε ότι θα άρετε τα εμπόδια, αλλά δεν θα τα άρετε αν με αυτά τα εμπόδια προστατεύονται τελικά οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές. Για τις ε, διοικητικές δυσκολίες. Φυσικά και πρέπει να εκτιμηθούν, να αξιολογηθούν και να δούμε τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για αυτά. Η Ευρωπαϊκή Αγορά δεν μπορεί να είναι ε, συνώνυμο ε, του ανταγωνισμού όσον αφορά τα ζητήματα κοινωνικής προστασίας. Επαναλαμβάνω, η ευρωπαϊκή αγορά δεν μπορεί να βάζει σε ανταγωνισμό τα κοινωνικά μας συστήματα. Μα τα κοινωνικά μας συστήματα είναι κάτι κεκτημένο, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, είναι και το ένα και το άλλο. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν και εγώ θα φροντίσω ώστε καμία χώρα μέλος να μην ε, τα χρησιμοποιεί για να στρεβλώνει τους κανόνες του ανταγωνισμού, μειώνοντας την κοινωνική προστασία. Και δεν είμαι αφελής. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι μπορεί να θέλουν κάποιοι να κάνουν, αλλά εγώ θα είμαι παρόν και υπεύθυνο με τα μέσα που θα έχω στη διάθεσή μου για να δω και να φροντίσω να διορθωθεί η κατάσταση. Και θα το κάνω, να ξέρετε. Ευχαριστούμε. Κρίστοφ Γκούντλερ, Renew. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε υποψήφι Επίτροπε, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας, πολύ πλούσια, πολύ πλήρης. Για 30 δευτερόλεπτα θέλω να επανέλθουμε στο μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που, όπω ξέρετε, είναι ένα φιλόδοξο εργαλείο το οποίο ανταποκρίνεται στο ερώτημα του πώ μπορούμε να δαπανίσουμε καλύτερα από κοινού. Σήμερα, ξέρετε, η έλλειψη ε, συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας και της ε, ασφάλειας κοστίζει, εκτιμάται, μεταξύ 25 ε, και 100 εκατομμυρίων ετησίων. Ετησίως. Χρειαζόμαστε αυτό το Ταμείο Άμυνα, το οποίο θα συντονίσει, θα ολοκληρώσει και θα αξιοποιήσει τι επενδύσει των κρατών μελών και θα τι μεγεθύνει. Με τη συνεργασία αυτή θα έχουμε μια καινοτόμο αμυντική βιομηχανία, ανταγωνιστική, στην οποία θα μπορούν να υπολογίζουν όλα τα κράτη-μέλη για τι αμυντικέ του επενδύσει. Πώ μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι θα αξιοποιηθεί αυτό το ταμείο με ε, τεχνολογίες εχμής και διαλειτουργικές κυρίως και σύγχρονες που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές επιχειρησιακές και στρατηγικές ανάγκες της Ευρώπης και των κρατών μελών της. Ευχαριστώ κύριε Μπρετόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρουγκλέρ το θέμα αυτό είναι ύψη τη σημασία. Το διατυπώσατε πολύ σωστά ω ερώτηση και ω προβληματική. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο. Το λέω ειλικρινά. Γιγάντιο. Αυτό που έγινε από το Κοινοβούλιο και την προηγούμενη Κομισιόν δεν ήταν κάτι δεδομένο. Όπως είπαμε, δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς. Η Ευρώπη πρέπει σήμερα να ξεκινήσει να εξοπλίζεται με δικά της αμυντικά μέσα. Αλλά η Ευρώπη έχει και τη δική της ιστορία και ξέρω πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα αυτό για πολλούς από εσάς. Καταφέραμε λοιπόν να βρούμε ένα μέσο, εξαιρετικά ευφυές θεωρώ, το οποίο προέκυψε χάρη στις προσπάθειες των βουλευτών, ε, των κ. Τόια και Κράσνοντέψκη, η δυνατότητα αφενός ε, δημιουργίας ε, κάποιε ομοσπονδίε, γιατί δεν αρκούν οι τεχνολογίε μόνο. Να συνδυαστούν λοιπόν ε, όλες μαζί οι χώρες ε, της Ευρώπης σε μια συμμαχία και το λέω πολύ ευθείας αυτά τα 13 δισεκατομμύρια ε, του Ταμείου για τα 7 επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν τεράστιο μοχλό ανάπτυξης όπως ξέρετε αλλά για κάθε πρόγραμμα τουλάχιστον τρει επιχειρήσει που θα προέρχονται από τρει διαφορετικέ χώρε. Οπότε σκοπό είναι να συνεργαστούν όλοι, να εμπλέκονται όλοι, διότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα, κυρίε και κύριοι, δεν είναι θέμα μερικών μεγάλων χωρών. Είναι θέμα που απασχολεί και αφορά όλους μας. Οπότε πρέπει να ξεκινήσει σταδιακά η ευαισθητοποίηση όλων. Αυτό το Ταμείο Άμυνα λοιπόν επιτελεί και αυτό το σκοπό. Ε, να, υπάρχει, ε, να φέρει αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμετέχουν όλες σε αυτό το πρόγραμμα, να υποφελούνται από αυτό όλες, γιατί αφενός έχουμε τις γνώσεις, τις ικανότητες και αφετέρου την ικανότητα να ευαισθητοποιηθούν όλες οι χώρες και να δημιουργηθεί μια λύση που θα ανταποκρίνεται στην προβληματική. Ε, αν έχετε μια συμπληρωματική ερώτηση και δεν έχω απαντήσει τα πάντα, θα σας απαντήσω ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ που μου το προτείνετε, δεν μπορώ να αρνηθώ τη συμπληρωματική ερώτηση, κάτι παραπάνω για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα, ε, τη διαστημική συνιστόσα. Το διάστημα είναι πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και τεχνολογιών ε, στη διαστημική τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων μας ε, και των ικανοτήτων μας στον τομέα της ασφάλειας. Ναι, λοιπόν, το Ταμείο για το Διάστημα υπάρχει με 16 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά αφορά κυρίως μη στρατιωτικέ ε, εφαρμογές Κοπέρνικος, Γαλιλαίου, Εγνός. Πώς θα μπορέσουμε ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του Ταμείου Άμυνας να αφιερωθεί πράγματι στην διαστημική βιομηχανία άμυνας. Θα είμαι σαφής, η διαστημική βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η δεύτερη ήπειρο στον κόσμο η Ευρώπη σε διαστημικά θέματα και θα παραμείνει. Αυτό είναι ουσιώδες για, ε, πολύ σημαντικό για την αυτονομία και την ανεξαρτησία μας. Αλλά η Ευρώπη έχει και μια συνιστόσα μη στρατιωτική, η οποία θα παραμείνει. Ωστόσο, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ε, διπλής χρήσης τεχνολογίας οι τεχνολογίε που θα χρησιμοποιήσουμε στο Ταμείο Άμενα, πολλέ από αυτέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο διαστημικό κλάδο με μη στρατιωτικέ εφαρμογές, αλλά και αν σκεφτεί κανεί τον τον Γαλιλαίο τώρα μα δίνει θέσει ε, με ακρίβεια εκατοστού και σύντομα χάρη στην εκβατική φυσική ε, θα μα δίνει ακρίβεια χιλιοστού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την προβολή δυνάμεων, ε, η ανθρωπιστικών διαδρόμων, μετά το έχουμε το Κοπέρνικους, με τις τεράστιες δυνατότητες ε, διεκπαιρέωσης δεδομένων που τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται για μη στρατιωτικούς σκοπούς, μερικές φορές για στρατιωτικούς σκοπούς. Εγώ θα είμαι υπέρ, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, αυτών των τεχνολογιών διπλής χρήσης ε, και στο δομέα του διαστήματος. Ευχαριστώ. Επόμενος, ο κύριος Εστεμπάν Κονζάλες Πόντς. Εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, Γιούρι. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε. Γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει ένας αναλογικός κόσμος και ένας ψηφιακός. Υπάρχει ένας κόσμος που μόνο ψηφιακός θα είναι στο μέλλον. Δεν υπάρχει έπειτα μια ε, ιδιότητα που να είναι μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Στο μέλλον θα είναι μόνο ψηφιακά όλα. Οπότε θα πρέπει και η Ευρώπη να είναι προσαρμοσμένη σε αυτόν τον ε, ψηφιακό κόσμο. Έπειτα να έχουμε ασφάλεια στην πνευματική ιδιοκτησία. Σίγουρα εμείς προχωράμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ρωτάω, πώς θα διασφαλίσετε αυτό το κατάλληλο πλαίσιο για την ψηφιακή εποχή και πώς θα προχωρήσετε με την έρευνα και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη, ώστε ακριβώς η Ευρώπη να μην αποτελέσει ψηφιακή απικία στο μέλλον των ΗΠΑ ή της Κίνας. Παρακαλώ κύριε Μπρετών. Ευχαριστώ, αξιότιμη Ευρωβουλευτά, για την ερώτησή σας. Για όλες, αλλά για αυτήν ζωτική σημασία, γιατί ε, ξέρουμε όλη τη συζήτηση που γίνεται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, συζήτηση και προβληματισμός που μας απασχολεί όλους. Πολλοί πολίτες φοβούνται. Και γι' αυτό η εκλεγμένη πρόεδρος ζήτησε μέσα στις πρώτες 100 μέρες να τοποθετηθούμε πολύ συγκεκριμένα για την ηθική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να καθησυχάσουμε. Και όπως κάναμε και με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, πρέπει να έχουμε δικέ μα κατευθυντήριε γραμμέ, γιατί είμαστε διαφορετικοί στην Ευρώπη. Η προστασία του ατόμου και η ηθική για μα στην Ευρώπη είναι σημαντικό. Θέλουμε να ξέρουμε τι βρίσκεται πίσω από του αλγόριθμου. Δεν λέω ότι τα υπόλοιπα δεν θα τα ρυθμίσουμε. Θα δούμε τι θα πει το σώμα. Εγώ θα το στηρίξω. Αλλά προς το παρόν. Δεν λέω ότι πρέπει όλα να τα ρυθμίσουμε, αλλά λέω ότι πρέπει να έχουμε μία συγκεκριμένη άποψη εμείς για αυτά τα θέματα. Γιατί τα 500 εκατομμύρια πολίτες μας το θέλουν και το ζητάνε αυτό. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι δεδομένα. Άρα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν τα δεδομένα τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα, υπάρχουν αυτά που δεν θέλουμε να δώσουμε και τα κρατάμε. Υπάρχει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης για τη βιομηχανία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Τα δεδομένα λοιπόν, οι υπολογισμοί και οι servers, οι οποίοι θα εκπαιδεύσουν τους αλγόριθμους και τέλος οι αλγόριθμοι. Οπότε, πρώτα απ' όλα, τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε μια πραγματική ε, πολιτική τεχνητής ε, νοημοσύνης είναι αυτό το τρίπτυχο. Δηλαδή να έχουμε δυνατότητες υπολογισμών και να έχουμε όλο και μεγαλύτερη ισχύ στην Ευρώπη και μετά οι αλγόριθμοι, αφού προηγουμένως τοποθετηθούμε βέβαια για το τι θέλουμε να κάνουμε. Και τώρα μπορείτε συμπληρωματική ερώτηση για να συνεχίσω, αν το επιθυμείτε. Κύριε Πόντς, συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, θα σας περιμένω και την επόμενη φορά που θα έρθετε εδώ. Πάντως, ε, σε ζήτησε η Επιτροπή να αρχίσει ο προβληματισμός για την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Κυριαρχία. Γιατί οι μεγάλες ε, επιχειρήσεις στον κόσμο δεν είναι ευρωπαϊκές. Αλλά η ψηφιακή κυριαρχία θα έρθει σε αντιπαράθεση με την ψηφιακή κυριαρχία των χωρών μελών το ίδιο και για την τεχνητή νοημοσύνη, που και αυτή θα έχει κάποια σύνορα. Οπότε ρωτώ, τι πιστεύετε για την ευρωπαϊκή ψηφιακή κυριαρχία εσείς και ποια είναι η γνώμη σας για τον ψηφιακό προστατευτισμό. Συγκεκριμένα, τι πιστεύετε για τον προστατευτισμό, πείτε μας. Είμαι κατά του προστατευτισμού, λέει ο κύριος Δεν είναι η λύση. Πρέπει να βρούμε διαφορετικές λύσεις και θα έρθω σε αυτό. Ε, μιλήσατε για τα δεδομένα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντιπρόεδρο που ήταν εδώ πριν και ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Προσπάθησα να βοηθήσω κι εγώ στην προηγούμενη ζωή μου. Συνεισέφερα κι εγώ ως Ευρωπαίος. Και θα θυμόσαστε ε, τον αγώνα που δώσαμε μαζί κύριε Πρόεδρε Τιμπού για όλα αυτά. Και έπειτα τον αγώνα που έδωσα με τον Τζιν Σέμπλερ που ήταν ο αντιπρόεδρος της ΞΕΠΕ και είπαμε σε όλες τις επιχειρήσεις προσοχή, προσοχή στα δεδομένα σας. Τα δεδομένα των Ευρωπαίων πρέπει να αποθηκεύονται, να τα επεξεργαζόμαστε λοιπά εδώ και να μην έχουν πρόσβαση άλλοι σε αυτά χωρίς εμείς να το ξέρουμε. Ολόκληρη εκστρατεία δώσαμε τότε. Τα δεδομένα λοιπόν, αφού με ρωτάτε, είναι η ζωή μου. Οπότε μπορείτε να είσαστε πεπισμένοι ότι θέλω μια Ευρώπη η οποία να ελέγχει τα δεδομένα της, να μπορεί να τα μοιράζεται με άλλους, αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια, κυρίως για την τεχνητή νοημοσύνη θα είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό και για το 4.0 και, και θα σταματήσω με αυτό, θα είμαι αδιάλακτος, θα είμαι μαζί σας, με την Επιτροπή σας, για να προβληματιστούμε για αυτά τα ζητήματα. Πιστεύω όμως ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα γιατί συμφωνούμε μεταξύ μας και αν χρειαστεί θα νομοθετήσουμε και από αυτό επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λέμπρετον. Κύριε Μπρετό, ο επόμενος είναι ο κύριος Τίμο Βολκέν εκ μέρους της Γιούρη για τους σοσιαλιστές. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, θα γίνεται υπερεπίτροπος εάν σας επιβεβαιώσουμε. Θα έχετε αρμοδιότητα για τον πολιτισμό, το διάστημα και την αμυντική πολιτική. Πώς θα κάνετε τη δουλειά σας με συνοχή και υψηλή ποιότητα με όλες αυτές τις γενικές διευθύνσεις. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Εγώ είμαι μέλος των σοσιαλιστών. Έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα για, όσον αφορά ηθικά ζητήματα ε, ενώπιον της Επιτροπής ε, πρόσφατα είχατε εκατομμύρια μετοχές ε, στην Άτος. Δεν είδαμε εμείς κάποια απόδειξη για την πώληση, πώς πωλήθηκαν, ε, που δόθηκαν. Ε, θα υπάρχουν άλλες απαιτήσει δικές σας προς την Άτος μετά η σύγκρουση συμφερόντων που ανέφεραν οι συναδελφοί δεν έχουν αποδειχθεί ε, σαφώς. Ο κώδικας διοντολογίας το λέει καθαρά. Εσείς αποσύρεστε και από ε, συμβάσεις ή δεν έχω καταλάβει κάτι καθαρά. Κύριε Μπρετό, ευχαριστώ για την ερώτησή σας κύριε Βουλευτή. Ε, ευχαριστώ. Είναι σημαντικές ερωτήσεις. Θα σας δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Το πρώτο που μου ρωτάτε είναι αν πράγματι εκχώρησα όλες τις συμμετοχές που κατήχα από την Άτος ε, και από όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Θεώρησα ότι ήταν καθήκον μου και το έπραξα. Έγινε πριν από αυτή την ακρόαση, επαναλαμβάνω, μέσω μιας ε, γαλλικής τράπεζας που γνωρίζουν πολλοί Γάλλοι, έχει πολλούς Γάλλους πελάτες και στην αγορά. Οπότε έχω εδώ στη διάθεσή σας μια βεβαίωση που αποδεικνύει ότι αυτό έγινε στην αγορά και σε κανένα μέλος της οικογένειάς μου. Θα αφήσω το αντίγραφο στην κυρία Πρόεδρο. Μπορεί να σα το διαβιβάσει αν το συζητήσετε. Είναι φυσιολογικό που μου το ζητάτε και πολύ φυσιολογικά σα δίνω αυτά στις βεβαίωσει. Είναι δημοκρατία και την σέβομαι. Ζητώ συγγνώμη αν δημιούργησα κάποια σύγχυση όπω είπατε. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν καθαρός. Το επαναλαμβάνω. Δεν θα παρασυρθώ πέραν ε, του κλάδου με τον οποίο θα είμαι επιφορτισμένο. Δεν έχω κανένα συμφέρον πλέον, το είπα, κύριε ε, Βόλκεν. Ε, για τις, τις επιχειρήσεις αυτές. Δεν έχουν κανένα συμφέρον σε αυτές τις επιχειρήσεις. Μηδέν. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν να παρασυρθώ ε, και να δράσω προς όφελος τομέα. Ίσως να μην σας αρέσω και να μην με επιβεβαιώσετε, αλλά αν αναλάβω θα, το αναλάβω τα καθήκοντά μου υπεύθυνα. Αντιθέτως, αν σε κάποια περίπτωση κάποια από τις επιχειρήσεις οι οποίες διεύθυνα έρθει ε, ε για να ελεγχθεί από μένα. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα πάει στον επίτροπο που θα πρέπει να λάβει την απόφαση εξ ονόματο τη Επιτροπή, χωρί εγώ να το αντιληφθώ. Και θα πω και κάτι παραπάνω. Αν για παράδειγμα υπάρχει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όπου η Άτο, για παράδειγμα, ε, θέλει να κάνει μια αγορά, ε, θα ζητήσω να φύγω από την αίθουσα. Δεν θα συμμετέχω στη συνεδρίαση. Γνωρίζω, κύριε Βουλευτά, του κανόνε τη διακυβέρνηση, του έχω εφαρμόσει όλη μου τη ζωή και θα εξακολουθήσω να του εφαρμόζω με την ίδια αυστηρότητα Προ όφελο των Ευρωπαίων, του γενικού συμφέροντο των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ κύριε Βόλκιν, έχετε ε, συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Μια απάντηση για τις ε, ε, για άλλες απαιτήσει που σας ζήτησα εξοδοτικέ. θεωρείτε ότι θα ήταν λογικό για τη βιομηχανία Ε, να ελεγχθούν τώρα αυτές οι βιομηχανίες οι ρυθμιζόμενες βιομηχανίες. Αυτό είναι για να έχουμε την, ε, ε, την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Ο συνάδελφός σας, ε, έκανε μια πρόοδο. Εκεί υπήρχε το πρόβλημα πιθανή σύγκρουση συμφέροντος και είπε ο ίδιος ότι φυσικά σε περίπτωση που χρειαζόταν για να ότι θα αποδείκνει την ανεξαρτησία του. Μην το πάρετε ω επίθεση προ εσά. Εμεί θα θέλαμε εσεί εδώ, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νομίζω ότι κατάλαβα αν τελειώσατε την ερώτησή σας. Ε? Τότε, αν μου επιτρέπετε, 10 δευτερόλεπτα έχω να τελειώσω με αυτά τα 10 δευτερόλεπτα την ερώτησή μου. Δώστε μου τη δυνατότητα να τελειώσω. Εγώ θέλω να τελειώσω την ερώτησή μου, αν δεν σας πειράζει να τελειώσω την ερώτησή μου. Λοιπόν, ο συνάδελφό σα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια πολύ επιθετική δήλωση. Εσεί μπορείτε αυτό να το κάνετε, το φαντάζεστε, όπου δηλαδή όταν θα έχετε θέματα που θα άπτονται τη άτο, εσεί ο ίδιο για να μην υπάρχει έστω και παραμικρή υποψία τη ε, σύγκρουση συμφερόντων με την άτο, θα αποσυρθείτε από μια τέτοια συζήτηση. Φυσικά. Πολύ καλή η σύστασή σα. Αυτό είχα σκοπό και να κάνω μάλιστα αλλά αφού με προκαλείτε να το πω, ε, ενώπιον σας αναλαμβάνω τη δέσμευση πράγματι σε καμία περίπτωση ποτέ δεν πρόκειται να λάβω να υποδεχθώ οποιοδήποτε μέλος της ε, επιχείρησης που εγώ διεύθυνα μόνος στο γραφείο μου βάσει του κώδικα διοντολογία για του επιτρόπου. Αυτό επιβάλλει όταν κάποιο υποδέχεται ε, λομπίστε, βιομηχάνου, δεν είναι ποτέ μόνο του. Ε, πρέπει να συνταχθεί και κάποια έκθεση. Είναι δημόσιε οι συναντήσει αυτέ. Η ατζέντα μου θα είναι δημόσια, το περιεχόμενο θα είναι δημόσιο, αλλά εγώ θα πάω και λίγο πιο πέρα. Σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια δυνατότητα θα ζητώ από κάποιον από τους επιτρόπους, ε, η κυρία Φεστάγκερ, ε, η, μια από τι δύο επιτρόπου, να είναι παρούσα ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία. Αμφιβολία για το πρόσωπό μου, γιατί είπα, το αναλαμβάνω σε ευθύνη ω επίτροπο, αλλά είναι πολύ καλή η σύστασή σα και δεσμεύομαι ενώπιον σα. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να υποδεχθώ μόνο μου μέλο μια επιχείρηση που διήθυνα στο γραφείο μου, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Μιλήσατε φυσικά για την σύνταξη. Ναι, έχω σύνταξη. Απλά είπα ότι αυτή η σύνταξη τώρα έχει εκαθαριστεί. Ε, ήταν μια μεγάλη ασφαλιστική επιχείρηση που θα μου την έδινε. Είπα ότι δεν θα την λαμβάνω όσο είμαι, δεν θα την εισπράττω όσο είμαι επίτροπο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν μπορώ να έχω μια απασχόληση ω επίτροπο και ταυτόχρονα να λαμβάνω κάποια σύνταξη. Θα την λάβω. Δεν έχει καμία σχέση με την Άτος. Εάν ε, η Άτος ε, χρεοκοπήσει. Ούτως ή άλλως εγώ θα λάβω τη σύνταξή μου, θα την εισπράξω κάποια στιγμή. Εγώ το ζήτησα, κανείς δεν μου το έχει επιβάλει, απλά είπα ότι θα την εισπράξω όταν θα φύγω από την Κομισιόν. Ελπίζω σε πέντε χρόνια, εάν μου δώσετε την εμπιστοσύνη σας. Uh, Επόμενη ερώτηση από τον κύριο Ράσμουσεν από τους ε, Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Μπρετόν το θέμα της ε, κυβερνοασφάλειας, συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη να προετοιμαστεί για την ψηφιακή εποχή. Και αναφερθήκατε ήδη στην οδηγία για το ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό εμπόριο, ε, το θέμα της ανάληψης ευθυνών, πολύ σημαντικό. Στις γραπτές απαντήσεις σας αναφέρετε νέους κανόνες για να στηρίξετε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Και τον Ιούλιο είπατε ότι είναι πιθανό με μονομένα άτομα στο μέλλον να πληρώνονται για δεδομένα. Άρα δηλαδή ένα σύστημα σύστημα όπου μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να προστατεύουν την ιδιωτική του σφαίρα. Πριν από λίγο είπατε ότι θα είσαστε ο Επίτροπος των Δεδομένων. Για μας τους πράσινους ε, ε, το θέμα της προστασίας δεδομένων είναι δικαίωμα των καταναλωτών και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Πώς μπορείτε λοιπόν να εξηγήσετε αυτά που είπατε στην αρχή του έτους για την προστασία των δεδομένων. Ως Επίτροπος θα πρέπει να προστατεύετε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές και για τα δεδομένα. Ε, γι' αυτό λοιπόν σας ε, ερωτώ, ε, σκοπεύετε να ενισχύσετε την βιωτική σφαίρα και την ασφάλεια όσον αφορά, παραδείγματος χάνει το θέμα των connected products. Πολλές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, από τις θέσεις στις οποίες βρέθηκα πάντα ήθελα να ευαισθητοποιήσω τους Ευρωπαίους συμπολίτε για το γεγονός ότι τα δεδομένα τους πρώτα απ' όλα ήταν δικά τους και δεύτερον ότι έχουν κάποια αξία. Και βλέπετε, έχω δει πολλά στη ζωή μου μέχρι τώρα. Ανθρώπους, επιχειρήσεις που δεν προσέχουν τα δεδομένα τους, ενώ είναι δικά τους, τους ανήκουν. Και αυτό θέλω να πω, αυτό είναι, έτσι πρέπει να καταλάβετε αυτά που λέω, ότι τα δεδομένα είναι δικά σας. Και πρέπει να μπορούμε να τα διαθέσουμε όπως θέλουμε. Φυσικά υπάρχουν και άλλα δεδομένα τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα. Και το υπενθύμησα και με τον πρόεδρο πριν, ότι και αυτό αποτελεί στοιχείο της Ευρώπης και είναι θεμελιώδου σημασία για την Ευρώπη. Σε αυτή την κοινή αγορά δεδομένων λοιπόν και ιδίω των βιομηχανικών δεδομένων υπάρχουν κάποια που είναι θεμελιώδου σημασία και οι επιχειρήσει θα θέλουν να τα κρατήσουν ε, για τι ίδιε, γιατί είναι πολύ σημαντικέ για την καινοτομία, την έρευνα κτλ. Και άλλα δεδομένα που θα πρέπει να τα μοιραζόμαστε μεταξύ μα, ανώνυμα ή όχι, ακριβώς για να μπορούν από αυτά να υποφεληθούν και άλλοι και η πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη. Άρα λοιπόν είναι διτό το ζήτημα. Προστασία και ελευθερία. Γι' αυτό και χρειάζεται ρύθμιση και γι' αυτό και στην Ήπειρό μας ρυθμίζουμε τα δεδομένα και θα συνεχίσω. Έπειτα μιλάτε για την ασφάλεια στο κυβερνοχώρο. Βεβαίω και είσαστε και εισηγητή για αυτό το θέμα και συγχαρητήρια για το έργο σας. Το παρακολούθησα και πριν έρθω εδώ. Πολύ σημαντικό για να ευαισθητοποιηθούν όλες οι επιχειρήσεις. Και ναι, είναι αλήθεια και πρέπει να τεθεί το ζήτημα της κυβερνοασφάλεια Και όταν ε, κατασκευάζουμε κάτι που μπορεί να είναι ζωτική σημασίας. Οπότε το θέμα της ε, ε, σύλληψης του μηχανισμού που μας προστατεύει στον κυβερνοχώρο είναι το πρώτο στοιχείο και μετά και η χρήση του βέβαια. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για μας μια πιο συγκεκριμένη απάντηση θα ήταν πολύ καλύτερη. Να σχολεία. Αυτά είχα να πω για την πρώτη σας ερώτηση. Απάντηση μάλλον. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι ότι εμείς ε, θέλουμε να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, ψηφιακή εποχή. Ε, εσείς έρχεστε από ψηφιακέ επιχειρήσεις στην Άτος, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία. Υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν κάποια προβλήματα στις τις απαντήσεις σας δώσατε κάποια στοιχεία. Είπατε ότι ε, δεν θα ε, έχετε καμία σχέση με οικονομικές αποφάσεις σε σχέση με την άτοση. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για τα οικονομικά, πρόκειται και για τις ε, ρυθμίσεις. Να μην επαναλάβω αυτά που είπαν οι άλλοι συνάδελφοι. Η Άτος δουλεύει για την κυβερνοασφάλεια, τηλεπικοινωνίες, την έρευνα για το διάστημα και σε πολλά άλλα θέματα. Θέλω να ακούσω από εσά τι είδου αποφάσεις πιστεύετε ότι έχουν σχέση με την βιομηχανία που θα αναλάβετε χωρίς να παρεμβαίνει η Άτος. Ως επίτροπος, τελικά τι μπορείτε να κάνετε ε, σε αυτό το χαρτοφυλάκιο χωρίς να έχετε καθόλου σε επαφή με την Άτος. Ο κύριος Μπρετό, καταλαβαίνω την ερώτησή σας και θα σας το ξαναπώ. Αναφερθήκατε διάφορους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Άτος και ευτυχώς δεν είναι και η μόνη επιχείρηση του κλάδου από τα 45 δις 0,1% επιδοτήσεις πήρε η Άτος τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 15 εκατομμύρια ούτε καν πέρυσι. Υπάρχουν πολλές άλλες επιχειρήσεις ε, του κλάδου και ευτυχώ. ναι, θα ασχοληθώ με όλες. Σας το είπα, δεν πρόκειται να ξεφύγω καθόλου. Όπως το έκανα και όταν έγινα υπουργός της γαλλικής κυβέρνησης. Και τότε στο χαρτοφυλάκιό μου είχα και τις τηλεπικοινωνίες, τους γνώρισα, από εκεί ερχόμουν, τους ρύθμισα όμως. Και χρησιμοποίησα ό,τι μέσα είχα στη διάθεσή μου για να πάω να ψάξω να βρω όπου υπάρχουν προβλήματα και ήμουν αδιάλακτος ως υπουργό. Δεν είναι επειδή προέρχομαι από ένα κλάδο που μπορεί να είναι ο ένας ή ο άλλος δεν μπορώ να κάνω και καλά τη δουλειά μου. Είμαι Γάλλος, δεν πρόκειται να ξεφύγω και να κάνω πως δεν καταλαβαίνω επειδή θα μιλάμε για τη Γαλλία. Όχι. Δεν έχω πλέον κανένα συμφέρον και το μόνο μου συμφέρον είναι το ευρωπαϊκό γενικό συμφέρον και αυτό θα κυριαρχήσει σε ολόκληρο το χαρτοφυλακιό μου. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Παύλο Μπόρκια από την Ήτρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς ε, προηγουμένως ε, αναφέρατε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άμυνα που αναφέρθηκε και σήμερα το πρωί σε διάφορες ε, απαντήσεις που δώσατε σε γραπτή μορφή. Πάντως, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, όταν ήταν υπουργό Άμυνα στη χώρα της, τότε ζητούσε τη δημιουργία αυτού του ταμείου. Και επιπλέον, εσείς επανειλημμένα προσκληθήκατε στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Ε, άρα δηλαδή η Ατό είχε πολλά ε, συμφέροντα με αυτό το ταμείο και άρα δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι δικαιολογημένε οι ανησυχίε που υπάρχουν ε, για, για το κατά πόσο θα είσαστε ουδέτερος. Ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η πλήρης πώληση ε, των μετοχών σας δεν αρκεί για να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει πλήρης διαχωρισμός ανάμεσα σε εσά ως ρυθμιστή και ως πρώην εκπρόσωπο αυτής της εταιρείας. 60 εκατομμύρια ευρώ πήρε η Άτος από το πρόγραμμα Horizon και σας ερωτώ, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να εγγυηθείτε την ε, ανεξαρτησία στην αξιολόγηση. Ε, πώς μπορείτε να το εγγυηθείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήσασταν και εσύ μέλος όλου αυτού πριν από λίγο καιρό. Και πώς θα εγγυηθείτε την ανεξαρτησία σας, την πλήρη ανεξαρτησία στη διαχείριση του Ταμείου της Άμυνας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπορκιά για τις ερωτήσεις σας. Επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω τι ρωτάτε. Έχετε δίκιο για τα νούμερα. Σας συγχαίρω πράγματι. Περίπου 60 εκατομμύρια έλαβαν οι επιχειρήσεις ε, εντός εξαιτίας. Ε, ως επιχορηγήσεις που κάθε φορά υπενθυμίζω ήταν διαγωνισμοί. Δεν ήταν δώρα. Γίνονται διαγωνισμοί, πρόσκληση για υποβολή προσφορών από υπηρεσίες, για υπηρεσίε και οι υπηρεσίε αυτέ έχουν καθημερινέ γραμμέ και αποφασίζουν να τα εκχωρήσουν. Υπενθυμίζω, μιλάμε για 500 προγράμματα, 45 εκατομμύρια ε, σε σχέση με τα 45 δισεκατομμύρια. Ε, καταλαβαίνετε, μιλάμε για 0,1%. Πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πήραν πολλά περισσότερα. Και πάλι αυτό δεν είναι λόγος που επαναλαμβάνω τέτοιες ερωτήσεις να με τίθενται όταν αυτές οι υπηρεσίες γίνονται βάσει διαγωνισμών, δεν έχουν σχέση με επιτρόπους, γίνονται βάσει κατευθυντήρων γραμμών πολύ συγκεκριμένων και μετά υπάρχει μια διαδικασία διαφανής και αυτή την εγγύηση σας δίνω και εγώ, διαφάνεια των δημοσίων διαγωνισμών. Το βλέπετε, όπως μπορείτε σήμερα, πώς έγιναν οι εκχωρήσεις, οι αναθέσεις. Όπως είπα, δεν είναι ο επίτροπος αυτός που το αποφασίζει επιστώ, την προσοχή σας, δεν αποφασίζει ο Επίτροπος. Υπάρχουν νομικοί κανόνες της Κομισιόν σε πλήρη διαφάνεια. Αλλά αν τεθεί οποιοδήποτε ερώτημα προς τον Επίτροπο, το είπα, εκείνη τη στιγμή δεν θα τεθεί σε μένα ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε υποψία. Ήθελα να το πω σαφώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επανέλθω σε αυτό, να το επαναλάβω και να το τονίσω ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Μπόρκια. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, όλες αυτές οι ερωτήσεις περί ακεραιότητας και ανεξαρτησίας ε, είναι φυσιολογικές. Τη στιγμή που η υποψηφιότητα, τα υποψηφιότητά σας πέρασε από την Νομική Επιτροπή με μία μόνο ψήφο διαφορά υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτοί εξετάζονται ε, εξονυχιστικά για να είναι σίγουρο ότι ε, πριν ξεκινήσουν τη δραστηριότητά του στο Κοινοβούλιο δεν έχουν αναπτύξει κάποια άλλα δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να είναι αντίθετη με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς ε, φύγατε από την Άτος μόλις πριν από λίγες εβδομάδες και διαρωτώ με. Αν είχαμε κάποιον υπάλληλο που τον εξετάζουμε για σύγκρουση συμφερόντων και πάνε, πάμε πίσω πέντε χρόνια. Εσείς πιστεύετε τώρα αυτές οι λίγες εβδομάδες που φύγατε φτάνουνε. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, με παθιάζουν τα ζητήματα περί διακυβέρνησης για τους υπαλλήλου του Κοινοβουλίου. Είναι πέντε χρόνια, για τους επιτρόπους είναι δέκα. Γιατί για μα η δήλωση συμφερόντων δεν είναι πενταετή, όπω συμβαίνει με του υπαλλήλου του Κοινοβουλίου, είναι δέκα χρόνια. Έχετε λοιπόν τη δήλωση συμφερόντων που υποβάλλεται στην Επιτροπή Γιούρη. Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι για τη διακυβέρνηση. Η Επιτροπή Γιούρη δεν ψήφισε όσον αφορά εμένα, αποφάσισε η Επιτροπή Γιούρη που είναι ανεξάρτητος φορέας, δεν ξέρω τι έγινε γιατί δεν είδα τα αποτελέσματα, αλλά αποφάσισε δημοκρατικά και ψηφίζοντα πράγματι ότι δεν υπήρχε ανάγκη να μου κάνουν συμπληρωματικέ ερωτήσει. Δεν ψήφισε για την ακαιρεότητά μου, για να δει αν ή όχι. Διαπίστωσε βάσει τη δήλωσή μου ότι δεν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων και ότι αν υπήρχαν επιπλέον ερωτήσει, υπήρξε μια προηγούμενο τι ρωτήσατε και έγινε συζήτηση. Χαίρομαι ε, που μπορώ να απαντήσω σε επιπλέον ερωτήσεις που μου τίθενται. Είναι η δημοκρατία, είναι φυσιολογικό. Κάτι τώρα περί διακυβέρνηση. Ακριβώς αυτό έκανε η Επιτροπή Γιούρη, όχι κάτι άλλο. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Ιζεμπέλα Ελένα Κλότς από το ECR για την Ήτρα. Κύριε Μπρετόν, βλέπουμε λοιπόν ότι έχετε ε, σε βάθος γνώσεις για τη βιομηχανία και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό θα είναι ένα κομμάτι του μελλοντικού σας ε, χαρτοφυλακίου. Εγώ θέλω να σας κάνω μια πιο λεπτομερή ερώτηση. Μια ερώτηση που αφορά σε πολύ σημαντικά βιομηχανικά θέματα. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σας σχετικά με το μέλλον του καταλόγου στρατηγικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα προϊόντα. Όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, αυτός ο κατάλογος έχει συσταθεί από το 2011 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως ε, το κομμάτι αυτό που θα ελέγχετε εσείς ε, ε, επικαιροποιεί αυτό τον κατάλογο κάθε τρία χρόνια. Άρα ε, θα υπάρξει επικαιροποίηση σύντομα. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η δική σας άποψη για το μέλλον αυτού του καταλόγου, αν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές σε αυτό τον κατάλογο στρατηγικών προϊόντων. Και θέλω να γνωρίζω και περισσότερα για το μέλλον αυτών των προϊόντων στην οικονομία, παραδείγματο χάρη για τον άνθρακα που είναι πολύ σημαντικός για την παραγωγή χάλιβα στην Ευρώπη. Ε, θα υπάρχει στον κατάλογο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι χωρίς ε, τον ε, το κάρβουν αυτό, δεν μπορούμε να παράγουμε χάλιβα. Εχθές είχαμε μία συζήτηση από αυτού και πρόκειται για το μέλλον 6 εκατομμυρίων εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια ερώτηση ζωτική σημασία αυτή, που όντω βρίσκεται στο κέντρο ε, των θεμάτων που εμένα με απασχολούν και των προτεραιοτήτων μου, εφόσον με επιβεβαιώσετε. Κοιτάξτε, η πρώτη ύλη είναι ζωτική σημασία και για την ενέργεια, αλλά και γενικότερα έχουμε όλη υπόψη μας το κοβάλτιο και άλλα συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για να πετύχει η βιομηχανική και τεχνολογική μας στρατηγική. Και εδώ είναι που θέλω να αναφερθώ στην ε, αλυσίδα αξιών και για την άμυνα και για την τεχνολογία και για την πράσινη βιομηχανία κτλ. Υπενθυμίζω ότι το 2017 δημοσιεύσαμε 27 κρίσιμες ε, τέτοιες, ε, συστατικά, κρίσιμα τέτοια συστατικά. Πρέπει να ενημερωθεί αυτός ο κατάλογος και να δούμε ποιες είναι οι προοπτικές που έχουμε. Γιατί όντως είναι θέμα κυριαρχίας, βιομηχανικής και τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης. Γιατί είναι αυτός ο χάρτης πορείας που μου έχει ανατεθεί για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό μου και γι' αυτό θα το προσέξω πολύ το θέμα. Νέα δημοσίευση το 2020, υπενθυμίζω, σε συνεργασία βέβαια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί πρέπει να συμφωνούμε όλοι, και βέβαια στρατηγικές για τους διάφορους κλάδους και διαφοροποίηση. Ίσως και δυνατότητα με ειδικά διορθωτικά ταμεία να δούμε μήπως στην Ευρώπη μπορέσουμε, γιατί ανακαλύπτουμε ε, τέτοιες ε, ουσίες και συστατικά και στην Ευρώπη, στο επέδαφός μας, αντί να τα φέρουμε από το εξωτερικό. Μήπως μπορέσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την ανάπτυξη αυτών των υλικών και μέσα στην Ευρώπη και την εξόριξή τους. Ευχαριστούμε. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντησή σας και για αυτά που είπατε, ότι πράγματι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Στις γραπτές σας απαντήσεις αναφέρεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Green Deal, ε, πρέπει να στηριχτεί ε, πράγματι έγινε πολύ σημαντική προτεραιότητα για το κοινοβούλιο μας. Συζητάμε για το θέμα αυτό διεξοδικά, αλλά όπως και σε πολλές άλλες αλλαγές ε, και αυτή η αλλαγή απαιτεί χρόνο και πολλά κονδύλια και ερωτώ κατά πόσον συμφωνείτε ότι το αέριο διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την αλλαγή, κυρίως σε σχέση με τη βιομηχανία και κατά πόσον πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, στηρίξει και να χρηματοδοτήσει υποδομές ε, αερίου κατά τα επόμενα έτη. Αυτή η απάντηση είναι πολύ σημαντική για να μπορούμε να αποφασίσουμε για να στηρίξουμε την υποψηφιότητά Σα Κύριε Μπρετόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας αυτή και θα απαντήσω στην τελευταία κυρίω παρατήρησή σας. Φυσικά και πρέπει στην Ευρώπη να έχουμε διαφοροποίηση όσον αφορά τον εφοδιασμό μας σε ενέργεια. Και εγώ πράγματι θα είμαι ο επίτροπος εκείνος ο οποίος δεν είμαι βέβαια αρμόδιος για την ενέργεια, έτσι. Από τη δική μου θέση και το χαρτοφυλακιό μου θα ε, προωθήσω τις ενεργειακές εκείνες μορφές που θα βοηθήσουν την ενεργειακή μας ανεξαρτησία. Δεν είμαι αφελής, ξέρω ότι διακυδεύεται με το φυσικό αέριο, ξέρω ποιοι είναι οι συσχετισμοί δυνάμεων και η γεωπολιτική, οπότε το επαναλαμβάνω, για την ανεξαρτησία της Ευρώπης πρέπει να υπάρχει και ενεργειακή ανεξαρτησία. Και για να υπάρχει αυτή σημαίνει διαφοροποίηση στον εφοδιασμό μας και μάλιστα και με πράσινη ενέργεια. Πραγματικά θα είμαι αυτός ο οποίος θα προσφέρει αυτό το αναγκαίο μείγμα που είναι αναγκαίο για την ε, ανεξαρτησία μας. Σας ευχαριστώ. Ε, ωραία. Ε, προχωράμε. Σαμπίν Πεχέιεν, ΕΛΚ, Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι τα μέσα ενημέρωση και τα οπτικοακουστικά μέσα ε, θα τύχουν τις ε, σημασίες που τους αξίζει, γιατί πρόκειται για ένα περίπλοκο θέμα, το πιο περίπλοκο ίσως που θα κληθείτε να ε, εξετάσετε. Και ποια θα είναι άραγε η πρώτη σας προτεραιότητα σε αυτόν τον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διτή μορφή αυτών των μέσων που ξεπερνάει απλά τα θέματα της αγοράς. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω αν προτίθεστε να συνεργαστείτε με τους άλλους αρμόδιους επιτρόπους Μαρία Γκαμπριέλ και κυρία Γιούροβα για να έχετε μια συνεπή πολιτική έναντι των μέσων ενημέρωσης. Θα με ενδιαφέρει να γνωρίζω ε, πάνω απ' όλα πώς προβλέπετε τη συνεργασία με την κυρία Γκαμπριέλ σε σχέση με το πρόγραμμα για την Ευρώπη και κατά πόσον σκοπεύετε να λάβετε υπόψη σας και το σκέλος των μέσων ενημέρωσης αλλά και το πολιτιστικό σκέλος αυτού του προγράμματος ο Μπρετόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φρέιεν. Ξέρω πόση δουλειά έχετε κάνει για τα ζητήματα αυτά. Ειδικότερα σου συγγήτρια. το είχαμε συζητήσει τότε τα οπτικοακουστικά μέσα. Ήταν πολύ σημαντικό και με την κυρία Κάμερα Βέρτε. Ήταν πολύ σημαντικό το θέμα είναι εξίσου σημαντικό οικονομικά και για την Ευρώπη, για την πρόοδο της Ευρώπης. Γιατί αυτή η πτυχή, αυτός ο κλάδος που, διακατέχεται, που χαρακτηρίζεται και από την ψηφιακή επανάσταση, σήμερα σαφώς βρίσκεται στο επίκεντρο των ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε στην Επιρώμα, μας για να διατηρηθεί η πολυμορφία, ε, η άνθηση των δημιουργών μας, ε, ε, η χρήση των νέων εργαλείων και ο ίσος ανταγωνισμός με τους ε, κολοσσούς. Ε, αυτή η ποσόστοση των ευρωπαϊκών έργων στις διάφορες πλατφόρμες ήταν καταπληκτικό επίτευγμα. Μπράβο σας. Πρόκειται για ένα σημαντικό διακύβευμα για τους Ευρωπαίους δημιουργούς. Γιατί λέω ότι είναι εξίσου σημαντικό, διότι περιέχει και ένα τεράστιο σκέλος κοινωνικό, αφορά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι λοιπόν αμεληταίο θέμα, είναι τεράστιο, σημαντικότατο, αλλά όπως και τα υπόλοιπα χαρακτηρίζεται από, θα έλεγα, την επίδραση της ψηφιακής, των ψηφιακών τεχνολογιών και του ρόλου της απουσίας διαμεσολαβητών που ε, χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες πλατφόρμες. Ε, οπότε, μέσω του προγράμματος Media και όλων των προγραμμάτων που θα μοιραστεί μεταξύ της κυρίας Γκαμπριέλ και μου, ε, το καλό είναι ότι γνωριζόμαστε καλά γιατί δουλεύουμε εδώ και καιρό μαζί. Αυτό έχει συμβεί και στην προηγούμενη επιτροπή, οπότε θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, αυτό σας δηλώνω εδώ και αυτή φυσικά με το δικό της σκέλος, εγώ με το δικό μου σκέλος για τα μέσα. Εμφανώς για να ε, δώσουμε τη δυνατότητα σε όλο αυτό το κλάδο να συνεχίσει να εξελίσσεται. Όπως είπα, να τον προστατεύσουμε, να τον μετασχηματίσουμε και να τον προβάλλουμε. Κυρία Φεργαΐν. Όπως ε, αναφέρατε ήδη, έχουμε την οδηγία για λεπτοκοστικό μέσα που τέθηκε πέρυσι ε, σε ισχύ και τώρα υιοθετείται από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μία από τις σημαντικότερες πράξεις της προηγούμενης ηττίας. Αυτή βασίζεται στο καθεστώς ε, ευθύνη ε, που ισχύει για τους παρόχους και για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό αποδείχθηκε αποτελεσματικό για τις τελευταίες δύο δεκαετίες και είναι σημαντικό για τις πλατφόρμες. Εσείς σε ποια θέση έχετε έχοντας κατά νου την επερχόμενη μεταρρύθμιση της οδηγίας οδηγίες περί ηλεκτρονικού εμπορίου και περί παροχής υπηρεσιών. Αναφέρεστε νομίζω στην ε, προσαρμογή στο Digital Services Act και στην προσαρμογή ενδεχομένω τη ε, οδηγία ε, ηλεκτρονικού εμπορίου του 2000. Όπω είπα, η ευθύνη των πλατφορμών και του περιεχομένου αναφέρεται σαφώ. Δεν υπάρχει γενική επιτήρηση, είναι σαφέ. Δεν αμφισβητούμε την αρχή τη προέλευση και προσαρμογή τη ευθύνη και εκεί φυσικά υπάρχουν υποχρεώσει και ευθύνε σε αυτέ τι πλατφόρμε. Έχει, σταματήσει, έχει αποφασιστεί αυτό και όπω είπα, θα υιοθετήσουμε την οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν την αλλάξουμε. Αν αυτή ήταν η ερώτησή σα, θα την προσαρμόσουμε προ την κατεύθυνση που είπα. Θα την περιγράψω σωστά και επίση ε, δεσμεύομαι ενώπιον σα να συστήσουμε ένα ε, σχέδιο δράσης για τα μέσα και τα οπτικοακουστικά μέσα. Θα συνεργαστούμε μάλιστα αν θέλετε, γιατί ξέρω ότι έχετε πολλές προτάσεις και ιδέες, πρέπει να υλοποιηθούν, να υλοποιηθούν τα, όλα όσα έχουν γίνει, παρένθεση για το περιεχόμενο του 30% πώς υπολογίζεται ανά λεπτό, ανά έργο, πρέπει να το συζητήσουμε, να αποφασίσουμε, ξέρετε ποια είναι η απόψή μου, επ' αυτού εγώ ήμουν υπέρ των λεπτών. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πιες Κάρλος, ε, Κάρλες Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρετό που ήρθατε. Έχω και εγώ ερωτήσεις. Πολλοί αναφέρθηκαν στο παρελθόν σας, δεν χρειάζεται να αναφερθώ και εγώ σε αυτό. Αλλά ρωτάω, πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να είναι κανείς υποψήφιος για επίτροπος όταν έχει ήδη περάσει αποθέσεις απουργού κτλ. Το να ασχοληθείτε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σήμερα, ενώ εσείς έχετε δημιουργήσει τη δικιά σας επιχείρηση και έχετε βοηθήσει πάρα πολλές, πιστεύετε ότι είναι ενοχλητικό να ασχοληθείτε με τα ψυχικά στην Ευρώπη, ενώ εσείς ο ίδιος είστε ένας από τους μεγάλους παίκτε στα ψηφιακά, το ίδιο και για την τεχνολογία. Όταν εσείς ήσασταν επικεφαλής μια ευρωπαϊκή επιχείρηση που αγωνίστηκε στις διεθνεί αγορές για να πετύχει αυτή την ευρωπαϊκή ε, τεχνολογική κυριαρχία. Θα μπορούσα να συνεχίσω, αλλά θα σταματήσω με αυτά. Κάτι άλλο όμω, ε, για το οποίο σας ακούμε λιγότερο, είναι για το περιβάλλον. Κάτι λίγο αγγίξατε, αλλά μια από τι μεγάλε προκλήσει που ανέφερε και η εκλεγμένη πρόεδρος Φοντερ Λάιεν είναι η πρόκληση κλιματική. Εσείς πώς θα συμπεριλάβετε στο χαρτοφυλάκιο σας την κλιματική αλλαγή και τι ρόλο πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει ο ευρωπαϊκός ψηφιακός κλάδος για να έχουμε μια πιο βόσιμη εσωτερική αγορά. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Βλέπετε, ακριβώς έτσι η εκλεγμένη πρόεδρος Φοντερ Λάιεν μου είπε να δεχτώ την πρότασή της δεδομένων όλων αυτών των κλάδων και των δομένων που έχω γνωρίσει στη σταδιοδρομία. Έχετε δίκιο. Η Πράσινη Συμφωνία θα είναι ζωτική σημασία. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι μάτια λόγια και ένα περιεχομένου. Όχι, πρόκειται για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στον κλάδο, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς. Πρόκειται για ένα όραμα για το 2050, έτσι, αλλά αύριο είναι το 2050. Όταν ε, θέλουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές ε, σε ένα εργοστάσιο, ας πούμε, να αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής, η αλλαγή, και το έχω ζήσει πολλές φορές στη ζωή μου, κάπου 25 χρόνια, βλέπετε, 25 με 50 Φτάσαμε στα 30. Λοιπόν, αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο του 2050, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις τα επόμενα 5 χρόνια για να γίνουν οι αλλαγές που χρειάζεται και να πετύχουμε τη φιλοδοξία μας το 2050. Άρα, αποτελεί μια κινητήριο δύναμη ε, τροποποίησης της βιομηχανίας μας. Εννοείται ότι θέλω μια ρύθμιση τομεακή, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, δράσεις. Ε, κυκλική οικονομία, νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα προϊόντα, όλα τα θέματα που έχουν για την ε, προγραμματισμένη φθορά και καταστροφή κάποιων ε, μηχανημάτων. Ενεργειακή μετάβαση, σας τα είπα, το αποτύπωμα άνθρακα που θέλουμε να καταργήσουμε. Και αυτό έχει να κάνει με τα ψηφιακά, γιατί ο ψηφιακός κλάδος δημιουργεί πάρα πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Άρα, πράγματι, βλέπετε ότι είναι ένας ολόκληρος βιομηχανικός κλάδος που θα προχωρήσει η βάση αυτής της φιλοδοξίας. Γι' αυτό και όλοι, τόσο μεγάλες επιχειρήσεις όσο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το όραμά μας για το 2050. Το τι θα γίνει τότε όμως θα παιχτεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Συμπληρωματική ερώτηση. Πολύ σωστά είπατε ότι η βιομηχανία πρέπει να πάει προς νέους ορίζοντες. Ναι, αλλά υπάρχει και ευθύνη των δημοσίων παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για πάρα πολλές υπηρεσίες. Υπάρχουν βέβαια στις δημόσιες προμήθειες ο περιβαλλοντικός παράγοντας στη διοντολογία και υπάρχει και η ευρωπαϊκή ρύθμιση πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά για να βελτιώσουμε συγχρόνως και την οικονομική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Και πιστεύετε ότι θα έπρεπε με τον ένα τον άλλο τρόπο, δεν ξέρω εγώ πώς, να βοηθήσουμε τις αρχές που χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά κριτήρια για να καταλήξουν σε απόφαση για τις δημόσιες προμηθειές τους. Και είναι πολλές οι αρχές που το κάνουν αυτό. Απάντηση. Ναι, έχετε δίκιο που το λέτε. Οι δημόσιες αγορές όντως αποτελεί έναν πάρα πολύ καλό μοχλό για να πετύχουμε το στόχο μας. Είναι το 80% του Και στις διάφορες προσφορές εγώ θα φροντίσω οι δίκτυες αυτοί, οι περιβαλλοντικοί, να ληφθούν υπόψη ε, κυρίως τη βαθμολόγηση για να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε κατά πόσο ένας ή ο άλλος υποψήφιος θα πάρει την προσφορά ή όχι. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει και ανταγωνισμός, να είναι ανταγωνιστική δηλαδή η προσφορά αυτή, έτσι, όχι μόνο περιβαλλοντική. Πάντως σήμερα παντω σημερα ότι δεν χρησιμοποιούμε του περιβαλλοντικού ε, παράγοντε και τα κριτήρια αρκετά. Αλλά θα το κάνω και θα κοιτάξω να σα συναντήσω για να δούμε μαζί πώ μπορούμε να το κάνουμε. Με μια ειδική ομάδα εργασία, ώστε να κινητοποιηθούν όλε οι κρατικέ αρχέ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δημόσιοι φορείς και θα διαπαιδαγωγήσουμε τον κόσμο προς αυτή την κατεύθυνση να λαμβάνουν υπόψη τους τα περιβαλλοντικά κριτήρια όταν αποφασίζουν για ε, τις δημόσιες προμήθειες. Ο κύριος Ιγνάθιο Κοράο, τώρα, Ήτρε, μη εγγεγραμμένος. Καλημέρα κύριε Πίτροπε κύριε Υποψήφιο επίτροπε. Έχω πολλού προβληματισμού όσον αφορά τι παλιότερε δραστηριότητέ σα. Υπάρχει υψηλό κίνδυνο σύγκρουση συμφερόντων. Ήθελα να σα ενημερώσω ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε και στην Κίνα μάχονται διαρκώ κατά για την τεχνολογική κυριαρχία παγκοσμίω. Η Ευρώπη φαίνεται να μην συμμετέχει στο μάτσα αυτό και εξαρτάται από του άλλου. Τώρα, επειδή αυτό που σας αναέθεσε η κυρία Βάντερ Λάιεν περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Ανεξαρτησία, ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να υιοθετήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά την έλλειψη μιας βιομηχανικής στρατηγικής. Κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις εξαγοράστηκαν από ξένους ομίλους ε, που μπλόκαραν την ευρωπαϊκή παραγωγή ή την μετέφεραν με σοβαρέ συνέπειε ε, στην ευρωπαϊκή ε, βιομηχανική ανεξαρτησία. Ένα παράδειγμα, ε, η χαλιβουργία στο Ταραντό. Τι θα κάνετε ε, στο πλαίσιο αυτού του Green, του New Deal, ε, για τη βιομηχανία, πώς θα χρησιμοποιήσετε την έρευνα και την κοινοτομία για βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη. Κύριε Μπρετόν. Ουσιαστικά πρέπει να το χτίσουμε όλο. Ευχαριστώ γιατί μου κάνετε ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένες Πράγματι, μέσω των ερωτήσεων σας αφενός έχουμε τη φιλοδοξία, στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως για το 2050 και μετά έχουμε τα κατεπήγοντα. Τα κατεπήγοντα, όπου ειδικότερα, ξέρουμε ότι υπάρχουν παντού, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις επικράτειες, όσον αφορά τη μετάβαση. Υπάρχουν εργαλεία φυσικά, τα οποία υπάρχουν και τα οποία θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε. Τα εργαλεία αυτά είναι τα ταμεία ε, μετάβασης ή ε, οικολογικής πράσινης, ε, πράσινου μετασχηματισμού. Θα είναι εργαλεία που θα μας εξοπλίσουν για να μπορέσουμε να παρεύουμε εκεί όπου μπορούμε και όπου πρέπει, ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη σημαντική μετάβαση την οποία ανέφερα προηγουμένως. Πέραν αυτού, εσείς αναφέρεστε, καταλαβαίνω την ερώτησή σας, όσον αφορά την ανάγκη αυτή να αρχίσουμε να ε, φτιάχνουμε ή να ενισχύσουμε τη βιομηχανική βάση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει ε, ε, στην Ευρώπη το 24% των θέσεων απασχόληση είναι αντιστοιχούν στη βιομηχανία και έχει να συναγωνιστεί παγκόσμιου ομίλου. Η βιομηχανία μα δεν είναι πρωταθλητή. Πρωταθλητέ μιλάμε είναι στο τέννη ή στο μπάσκετ. Είναι ε, κάτι άλλο η βιομηχανία και Χρειαζόμαστε μεγάλες βιομηχανίες για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε εισάξια στο παγκόσμιο ε, στερεώμα. Γιατί χρειάζονται μεγάλες ε, επιχειρήσεις ε, για να μας παρέχουν δυνατότητες έρευνας και κοινοτομίας αλλά και για να υπάρχουν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μεγάλων επιχειρήσεων που θα συναγωνίζονται τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ε, από τι ΕΠΑ και την Κίνα και εγώ από τη θέση μου θα κάνω τις σχετικές προσπάθειες ε, φυσικά στην συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο ε, και την συναδελφό μου την κυρία Μάγκρετ Φεστάγκερ. Ευχαριστούμε κύριε Κοράου. Συμπληρωματική ερώτηση, ναι. Δεν κατάλαβα πολύ καλά τι μέτρα ακριβώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθεί αυτό το κενό τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας είτε αν μιλάμε γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα ε, σε θέματα τεχνολογικής, ε, ε, τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με τη ΣΥΠΑ ή την Κίνα. Και τώρα για την άλλη ερώτηση, όσον αφορά τα βιομηχανικά σχέδια σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Green Deal, δεν καταλαβαίνω με ποια εργαλεία σκοπεύετε να γίνεται ο μετασχηματισμός. ή να υποστηρίξετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λόγω του κόστου των πρώτων υλών ε, και άλλων ε, κανόνων που υπάρχουν συχνά παραμένουν στο περιθώριο. Θέλω να μου πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Τι είδους δράσεις σκοπεύετε να υλοποιήσετε. Ευχαριστούμε κύριε Μπρετού. Ε, κύριε Βουλευτά, για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω υπάρχουν ταμεία κονδύλια τα οποία υπάρχουν για να βοηθήσουμε σε αυτή τη μετάβαση. Σε αυτές τις μεταβάσεις θα τα χρησιμοποιούμε η Κομισιόν θα επικεντρωθεί στο να μάθει πώς να τα αξιοποιήσει στο μέγιστο. Ε, στο νόμο έχω τώρα το Ταμείο Συνοχής ε, φυσικά, αλλά όπως είπα, με αυτό το Ταμείο Συνοχής ε, σε κάθε, ε, ε κάθε κράτος θα αποφασίζει την επενδυτική στρατηγική που θεωρείται είναι καταλληλότερη κατά περίπτωση. Εσείς αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν έχουμε χάσει τη μάχη, ούτε τον πόλεμο. Το είπα και προηγουμένω. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι δεδομένα, ε, υπολογιστική δύναμη και αλγόριθμοι. Τα δεδομένα δημιουργούνται διαρκώ. Δεν σταματάει αυτό σήμερα. Όλο ο πλανήτη είναι 40 τεραμπάιτ δεδομένα. Σε 5 χρόνια θα είναι 175 ε, τεραμπάιτ. Ε, τετραπλάσια δηλαδή. Δημιουργούμε αυτά τα δεδομένα. Το θέμα είναι να τα έχουμε ε, στη διάθεσή μας, να υπάρχει ο όγκος δηλαδή και να τα κατευθύνουμε σωστά προς να τα δρομολογήσουμε προ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει τη βιομηχανία μα με αλγόριθμου που να λειτουργούν καλά. Δεν έχουμε χάσει τον πόλεμο όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με του Αμερικανού και του Κινέζου. Σα το υπόσχομαι και θα είμαι παρόν με, με όλου ε, που θα με συνοδεύσουν σε αυτή τη μάχη σε όλε τι γωνιές του πλανήτη. Είμαι πεπισμένο, βαθιά πεπισμένο. Ευχαριστούμε ο κύριος Κάρλο Καλέντα από την Ήτρε, επόμενος εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Ε, πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο που έχουμε έναν υποψήφιο επίτροπο ο οποίος έχει μια ουσιαστική εμπειρία από επιχειρήσεις. Γιατί ο ε, άνθρωπος αυτός δεν θα ασχοληθεί με ψάρια αλλά με επιχειρήσεις. Άρα δηλαδή έχουμε τουλάχιστον ένα, ο οποίος ολόκληρη τη ζωή του δεν ήταν ε, πολιτικός και να μην λέμε τώρα ότι αυτός δεν μπορεί να έρθει σε υψηλά αξιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό θα ήταν ένα τεράστιο λάθος. Ε, αυτών λεχθέντων. Εκεί που εγώ ανησυχώ είναι ε, το θέμα της διάστασης απόψεων, ουσιαστική διάσταση απόψεων με την κυρία Βεστάγκερ όσον αφορά τις, ε, τις, τα, τις εθνικές νομοθεσίες, εθνικές, ε, τους εθνικούς πρωταθλητές. Νομίζω ότι λέτε αυτό είναι κάτι πολύ δυσάρεστο. Ε, δεν είναι καλό να προβάλλουμε αυτό έναντι των κρατών μας. Δεν ξέρω, πώς μπορείτε λιγάκι να το διευκρινίσετε. Δεν είναι... Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας και τα σχόλιά σας. Τα οποία προσωπικά συμμερίζομαι, εννοείται. Θα σας ε, εκπλήξω όμως για δεύτερη φορά, γιατί ε, δείχνετε, φαίνεται να λέτε ότι έχω διάσταση απόψεων με την αντιπρόεδρο Φεστάγκερ. Για το θέμα της Siemens, ξεκάθαρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε άλλη δυνατότητα από το να υιοθετήσει την απόφαση που υιοθέτησε σύμφωνα με τους κανόνες και αυτό έκανε. Το ζήτημα που τίθεται και έθεσε η εκλεγμένη πρόεδρος η κυρία Φοντερ Λάιεν τέθηκε δημόσια. Είναι ότι να δούμε και άλλα πράγματα, το συσχετισμό δυνάμεων και το πώς τα ψηφιακά επηρεάζουν την κατάσταση και τι αντίκτυπο έχουν τη στιγμή που τα έχουμε σε όλο το φάσμα. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοστούν όλες οι πολιτικές μας τις εξελίξεις. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε ε, την Ήπειρο με πολιτικές που υιοθετήσαμε πριν από 25 χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό. Μα ζήτησαν λοιπόν να το ξανανοίξουμε το ζήτημα και εγώ θα συνεισφέρω προς αυτή την κατεύθυνση. Θα το κάνω. Ε, αγορές ε, στα ψηφιακά δεν είναι όπως ήταν πριν από 25 χρόνια. Τότε δεν είχαμε τις πλατφόρμες, ούτε καν πριν 15 χρόνια. Τι σημαίνει ε, καλές, σωστές αγορές. Το θέτω, εντάξει, αφελώς, όχι αφελώς. Γι' αυτό λέω ότι θα είμαι αποφασισμένος για να γίνει αυτή η δουλειά που μου ζητήθηκε και θα είμαι πάντα πιστός στις αρχές. κύριος Καλέντα, για συμπληρωματική ερώτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, δεν εκπλήσωμαι. Ε, δεν με βάση αυτά που έχετε πει κατά παρελθόν. Λαμβάνω υπόψη, βέβαια, υπόψη μου ότι αυτή είναι μια δικαιολογημένη αλλαγή. Και θέλω να πω και το εξή. Αν τελικά είναι απαραίτητο να υπάρχουν ε, Ευρωπαίοι πρωταθλητές εισαγωγικά. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν. Αυτός ο κίνδυνος του να υπάρξει συγκέντρωση στην αγορά όχι μόνο για τους ε, καταναλωτές αλλά και για τους ε, παρόχους ε, που συνήθως είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους στρατηγικού τομείς όπως είναι το μέσο τη Άμυνα, Κατά την άποψή σα τι ακριβώ γραμμή πρέπει να ακολουθήσουμε σχετικά με το θέμα αυτό. Κύριο Μπρετό. Είμαι υπέρ του ανταγωνισμού. Είμαι υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισμού. Είναι μια αξία πάνω στην οποία δημιουργήθηκε η ενιαία μας αγορά. Είμαι φανατικός του ελεύθερου ανταγωνισμού και κατά των μονοπωλίων, ε, κατά των ε, εισοδηματιών. Αλλά το λέω ότι πρέπει να ξανανοίξουν κάποιες υποθέσεις. Μεταξύ άλλων, και ευχαριστώ που το θέσατε κύριε Καλέντα, όχι μόνο να δούμε τις επιπτώσεις της επιχειρήσεις, αλλά να δούμε και το σύνολο του οικοσυστήματος. Πια δεν είμαστε ένας κλειστός κύκλος. Η επιχείρηση πια είναι μια λυσίδα. Και έχετε δίκιο. Και το βλέπω και από την ερώτησή σας τι έχετε στο μυαλό σας. Επειδή θα έχουμε μεγάλους βιομηχανικούς συνασπισμούς, θα αναγκαστούμε να φέρουμε μαζί μας και ολόκληρες αλυσίδες ε, προμηθευτών. Αλλά αυτό το έχω ζήσει κι εγώ στη ζωή μου. Δεν είναι γεωγραφικά περιορισμένο αυτό το φαινόμενο, είναι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ευχαριστούμε κύριε Μπρετό. Τώρα θα δώσω το λόγο στο συνάδελφό μου, τον κύριο Γκρεζοντεύσκη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε τώρα τις τελευταίες έξι ερωτήσεις. Ο πρώτος των τελευταίων έξι είναι ο κύριος Μάντερς από το ΕΛΚ, ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κύριε Υποψήφιε, ε, θέλουμε να ενισχύσουμε, την, να στηρίξουμε την κοινή αγορά, αλλά ε, αυτό είναι πολύ χρονοβόρο το 80% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, δραστηριοποιούνται μόνο στη χώρα τους ε, γιατί υπάρχουν ε, δυσκολίες στο να εφαρμόσουν διάφορες οδηγίες. Εμείς θέλουμε να επιτύχουμε πλήρη εναρμόνιση, σαφείς κανόνες και επίσης θέλουμε και να έχουμε πιο σύντομες ε, διαδικασίες σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, γιατί όλα αυτά είναι πολύ χρονοβόρα. Παράδειγμα, το 2009 καταθέσαμε μία τροπολογία για να υπάρχει ο ίδιος φορτιστής για μικρά κινητά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ομόφωνα το ενέκριναν και τώρα όμως φτάσαμε στο 2019 ε, μετά από 10 χρόνια και ήρθε η Επιτροπή και πάλι με μία μελέτη που αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει, να γίνει έρευνα σε αυτόν τον ε, ε, φορτιστή, που, τον, ενιαίο, τον κοινό φορτιστή. Εκνευρίστηκαν όλοι γιατί περάσανε 10 χρόνια. Φαίνεται λοιπόν ότι μια τεράστια εταιρεία είναι εκείνη που θέλει να υπάρξει αυτή η αναβολή και εξακολουθούμε να έχουμε 51 εκατομμύρια τόνους ε, αποβλήτων κάθε χρόνο ε, γιατί σήμερα τα κινητά είναι πολύ σημαντικά για την καθημερινή μας ζωή. Άρα δηλαδή είναι απαραίτητο να φορτώνει κανείς την μπαταρία του κινητού. Και έτσι, ε, μισό λεπτό, ε, τι θα κάνατε λοιπόν αν εσείς τότε ήσασταν επίτροπος κοινή αγοράς. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι θέλετε να αποφασίσετε για νέα πρότυπα για ε, Wi-Fi συνδέσεις και τι θα κάνετε για να εναρμονιστεί η νομοθεσία. Δεν θα κάνετε ερώτηση μετά follow-up, τα δύο σας λεπτά τα φάγατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε. Χαρακτηριστικό το θέμα αυτό των όσων πρέπει να γίνουν και ευχαριστώ που το αναφέρατε διότι αφορά πολλούς συμπολίτε μας. Πρώτα απ' όλα να πω έγιναν κάποια πράγματα. Μου λέτε τι θα, έκανα, είχα κάνει εγώ. Αυτοί που προηγήθηκαν εμώ έκαναν πολλά. Ε, ε, εθελοντικά φυσικά γιατί η προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν προαιρετική αλλά μείωσε τον κατακρεματισμό. Ξέρω ότι ε, δεν έγιναν τα πάντα. Το 2018 η Κομισιόν ζήτησε από τον κλάδο να καταλήξει μια συμφωνία προαιρετική αλλά συμφωνώ μαζί σας εγώ είμαι νέο εδώ, ξέρετε. Μόλι ήρθα. Εγώ θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνεται στι απαιτήσει των καταναλωτών. Συμφωνώ μαζί σα. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα έχουμε μια εκτίμηση αντικτύπου που έχει ξεκινήσει ε, βάσει μια μελέτη, γιατί η προηγούμενη επιτροπή δεν έμεινε ικανοποιημένη. Εγώ θα την επιταχύνω. Μήπω καταλήξουμε και σε κάποια νομοθετική πρόταση. Θα δούμε ε, την εκτίμηση αντικτύπου λοιπόν για να επαληθεύσουμε τι συμβαίνει και ε, στην ανάλυση αντικτύπου θα δούμε ποιε ήταν οι επιπτώσει για του καταναλωτέ, τη βιομηχανία, το περιβάλλον και τι πιθανέ καινοτομίε μπορούμε να έχουμε. Ευχαριστώ την προσοχή σα στι καινοτομίε γιατί ενίο φορτιστή θα επιτρέπει. Ξέρουμε, ε, θα βασιστεί σε σημαντικέ τεχνολογικέ καινοτομίε. Αν είναι μια ε, νέα ενίο φορτιστή, θα περιλαμβάνει πολλέ τεχνολογίε και μπορεί να είναι και μεγάλο σε μέγεθο. Δεν είναι μόνο θέμα προτύπων και στάνταρ και δεν είναι κάτι εύκολο αλλά σας το λέω καθαρά αφού με ρωτάτε καθαρά και σας πήρε ώρα μάλιστα για να τη διευκρινίσετε. Εάν δούμε ότι η εκτίμηση αντικτύπου δεν δίνεται επιθυμητά αποτελέσματα, σας το λέω σήμερα, τότε θα θεωρήσω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προτείνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία βάσει τη συνήθους ε, ε, ε, νομοθετική διαδικασία. Θα το δούμε δηλαδή. Και αν δεν μείνουμε ικανοποιημένοι, θα κινηθούμε προς τα εκεί που λέτε εσεί. Έχετε ένα λεπτό ακόμα κύριε Μπρετό αν θέλετε. Κύριε Μάντερ, έχετε ένα λεπτό ακόμα. Όχι, εσείς δεν έχετε, γιατί το φάγατε το χρόνο σας προηγουμένως. Τα... Φάγατε τα δύο λεπτά που είχατε. Ο κύριος Μπρετόν έχει ένα λεπτό στη διάθεσή του. Αυτή είναι μια απόφαση του Πρόεδρου. Κύριε Μπρετόν, άμα θέλετε να μιλήσετε για άλλο ένα λεπτό. Νομίζω ότι χρησιμοποίησα το χρόνο μου, τον εξάντλησα, δεν χρειάζεται άλλο. Επόμενο ομιλητή είναι η κυρία Κονέτσνα, Ήμκο ε, και ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Εκτός από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ε, νομικά, μια νομική βάση ε, και μπορέσατε να μας ε, διαιρέσετε και να δημιουργήσετε διχασμό ανάμεσα σε πολλούς οργανισμούς. Θέλετε να δαπανίσετε τα χρήματα, αλλά το 10% του αμυντικού ταμείου θα πρέπει να κατευθυνθεί σε ρηξικέλευτες τεχνολογίες η εταιρεία στην οποία δουλεύατε είναι κορυφαία. Υπάρχουν επίσης πολλές άλλες χιλιάδες εταιρείε σε το τομέα. Εσείς δουλεύατε για μια εταιρεία που ήταν κυρίαρχη στον εφοδιασμό της, ε, στις προμήθειες που στην γαλλική κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι ε, πέρα από το να μην ανακατεύεστε σε αποφάσεις για συμβάσεις, για ε, επιλογές, μήπως ε, θα ήταν καλύτερα να παρετηθείτε και από τη θέση του Γενικού Διευθυντή για θέματα άμυνας, γιατί πάντα θα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Κοιτάξτε, είπα αυτό που ήθελα, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό, επαναλαμβάνω, να καταλάβουμε καλά στη, σε θέματα διακυβέρνηση αυτό που είπα προηγουμένω. Το υπενθύμησε και ένα βουλευτή ε, πριν λίγο. Έχω εργαστεί στη ζωή μου σε πολλέ επιχειρήσει. Σε υπουργεία, σε περιφέρειε. Και ξέρω πώ πώς να είμαι ανεξάρτητος. Δεν είναι επειδή ήμουν υπουργό Γάλλο που θα ευνοήσω τη Γαλλία. Ε, ως βουλευτής ε, ε, δεν εξυπηρετώ μόνο τον τόπο που γεννήθηκα, αλλά το γενικό συμφέρον. Όταν είμαι επίτροπος λοιπόν δεν ευνοώ τη χώρα μου. Λοιπόν, το ότι θα είμαι Γάλλος επίτροπος δεν θα σημαίνει ότι θα ευνοώ τη Γαλλία. Επειδή εγώ ε, δημιούργησα το Futuroscope που ήταν το πρώτο τουριστικό, θεματικό τουριστικό πάρκο στην Ευρώπη, δεν πρόκειται να ευνοήσω τον τουρισμό. Γι' αυτό τον λόγο επειδή η επιχείρηση που μόλι εγκατέλειψα ε, εργάστηκε πολύ λίγο από ό,τι πιστεύετε στον τομέα τη άμυνα, δεν σημαίνει αυτό ότι θα υπερασπίζω την άμυνα. Οι κανόνε διακυβέρνηση είναι σαφεί και θα του ε, εφαρμόζω αυστηρά. Τώρα, επί τη ουσία, η συνοχή στο χαρτοφυλάκιό μου περιλαμβάνει και αυτή τη νέα Γενική Διεύθυνση που θα συσταθεί, δεν έχει ακόμη συσταθεί και που θα έχει του στόχου τη. Ε. ε, θα είναι η Γενική Διεύθυνση Άμυνα και Διαστήματο. Είναι ουσιώδου σημασία γιατί η προστασία αυτού του τέταρτου διαστήματο που ανέφερε, το τέταρτου χώρου που είναι ε, οι πληροφορίε, ε, επίση ε, ε, περιλαμβάνει πολλέ πτυχέ που θα πρέπει να μα προβληματίσουν και να συνεργαστούμε. Και εδώ στο Κοινοβούλιο θα έρχομαι εδώ συστηματικά για να σα εξηγώ πώ θα χρησιμοποιούμε όλε αυτέ τι λειτουργίε, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την άμυνα στον κυβερνοχώρο, όλε αυτέ οι πτυχέ που ανέφερα προηγουμένως ε, χαρακτηρίζονται σήμερα από τις πτυχές του διαστήματος ε, και της άμυνας. Είναι, ε, χαρακτηρίζεται από συνοχή λοιπόν το χαρτοφυλάκιο, γι' αυτό έχει δημιουργηθεί έτσι. Ελπίζω να με επιβεβαιώσετε ως Επιτρόπο για να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε, διότι δεν έχουμε να χάνουμε ούτε λεπτό. συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ. Ωραία. Άρα δηλαδή εσείς θα εφαρμόσετε το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πρόγραμμα, παρότι σας λέω ότι αντιβαίνει στο πνεύμα της ιδρυτικής συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος πάντων, αν πρόκειται λοιπόν να τα εφαρμόσετε όλα αυτά, εγώ έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, ε, να προσφέρετε ως ε, εγγύηση ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να ξέρω πολύ συγκεκριμένα τι ελέγχους θα μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν θα πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα η εγγύηση και να το πω σαφώς είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για αυτό το ταμείο έχουμε την εγγύηση ότι τα επενδυτικά σχέδια θα παρουσιάζονται και θα συζητώνται στο Κοινοβούλιο. Έτσι δημιουργήθηκε το Ταμείο. Και φυσικά και θα το πράττω και σίγουρα περισσότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά. Συγγνώμη που επανέρχομαι, αλλά και εδώ επαναλαμβάνω, διακυβέρνηση, δίκαιο είναι κάτι σημαντικό. Ξέρω ότι κάποιοι συζήτησαν ε, επειδή, το, για το κατά πόσο νομιμοποιείται η δημιουργία ενό τέτοιου ταμείου. Το άρθρο 41.2 αναφέρεται σε επιχειρήσει και απαγορεύεται στην Ένωση να χρηματοδοτήσει επιχειρήσει στρατιωτικέ. Αλλά η νομική βάση, όπω το γνωρίζετε, γιατί συζητήθηκε εκτενώ στο Κοινοβούλιο εδώ, η νομική βάση επί τη οποία ε, βασίζεται η νομοποίηση του Ταμείου, το οποίο δεν είναι παράνομο, το είδαν όλε οι νομικέ υπηρεσίε. Είναι το άρθρο 173 και αφορά τι βιομηχανικέ πτυχέ και το άρθρο 186 που αφορά την έρευνα. Το επαναλαμβάνω γιατί και εγώ εξέτασα με μεγάλη ε, προσήλωση αυτό το ζήτημα. Ξέρω ότι συζητήθηκε πολύ. Ήθελα να σχηματίσω και εγώ γνώμη και σα επιβεβαιώνω ότι το υποστηρίζω 100%. Ευχαριστούμε. επόμενο ομιλητή είναι ο κύριος Μπενιφέη, ΙΜΚΟ, ε, Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, υποψήφιοι Επίτροπε, κύριε Μπρετόν. Ε, αυτή τη στιγμή ε, κάθε πέμπτος ε, Ευρωπαίος πολίτης έχει ένα, ε, μια συσκευή smart, άρα δηλαδή μιλάμε, θα προκύψουν όλο και περισσότερες αλλαγές και προκλήσεις. Εσύ μας είπατε ότι η τεχνητή νομοσύνη βασίζεται σε δεδομένα και σκοπεύετε να έχετε κοινό ευρωπαϊκό χώρο για τα δεδομένα. Σας ερωτώ λοιπόν, πώς θα εγγυηθείτε ότι κάθε νομική πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη θα δεν θα φέρει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι η ιδιωτική σφαίρα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, ποια είναι μια καλή και ουσιαστική ευρωπαϊκή προοπτική και ποια είναι η στρατηγική σας ε, για την τεχνητή νομοσύνη. Ε, υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών. Σας ερωτώ λοιπόν, τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην χρησιμοποιείται με διακριτική μεταχείριση βάρος ανθρώπων όσον αφορά ας πούμε την υγεία τους, την εθνοτική τους προέλευση, την προσωπική τους κατάσταση, γιατί ελοχεύει σαφώς αυτός ο συγκεκριμένος κίνδυνος. Κύριε παρακαλώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας υπενθυμίσω ότι η σχέση μας με όλα αυτά τα ερωτήματα βασίζεται στην οδηγία του 2000 για το εμπόριο. Μην ξεχνάμε τα βασικά. Τα βασικά αυτά στοιχεία δεν θα αλλάξουν τα θεμέλια. Σας το επιβεβαιώνω. Σας ε, διαβεβαιώνω. Ε, αφορούν την προσέγγιση μας προς τα δεδομένα. Θα επανέλθω σε κάποια βασικά στοιχεία που δεν πρέπει να ξεχνάμε καμία γενική επιτήρηση, εποπτεία, καμία αρχή ε, χώρας προέλευσης και προφανώς ευθύνη για τις μεγάλες πλατφόρμες, που θα έχουν οι μεγάλες πλατφόρμες να ε, επιβλέπουν ώστε όλοι οι παρεμβαίνοντες, όσοι θα δραστηριοποιούνται σε αυτό το περιβάλλον δεδομένων, να τηρούν τα θεμελιώδη στοιχεία, όπως τα έχουμε ορίσει εμείς. Ε, να αποφεύγονται οτιδήποτε αφορά το μίσος, τη διακριτική μεταχείριση, την τρομοκρατία, όλα τα μηνύματα ε, που έχουν χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας και και όλα τα σχετικά υπάρχουν κανόνες και πρέπει να του προσαρμόσουμε επαναλαμβάνω αλλά για άλλη μια φορά η ελευθερία που είναι εγγενής στον κόσμο των δεδομένων για μένα είναι θεμελιώδη ελευθερία πρέπει να διατηρηθεί θα διατηρηθεί. Σας το επιβεβαιώνω ότι πράγματι με αυτή τη λογική σκέφτομαι. Ε, κατά τα άλλα, μάλιστα, διαφέρουμε από τις άλλες μεγάλες υπήρους. Η ιδιαιτερότητά μας, η γνησιότητά μας, η αυθεντικότητά μας ε, και να πω και κάτι παραπάνω, όσα καταφέραμε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ε, δημιουργώντας, ελπίζω, σύντομα ένα παγκόσμιο πρότυπο, Πιστεύω ότι ο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα και αυτό που αναφέρατε προηγουμένω, που αφορά του κανόνε ηθική που θα αρχίσουμε να ορίζουμε για τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη μέσα στι 100 επόμενε μέρε, θα πρέπει να αποτελέσουν σημείο αναφορά και για εμά, του Ευρωπαίου πολίτε, και για τον υπόλοιπο κόσμο ενδεχομένω. Συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο συνδεδεμένο θέμα, γιατί η συνεργατική οικονομία, η collaborative economy, έχει σχέση και με την τεχνητή νομοσύνη και στις γραπτές σας απαντήσεις είπατε ότι αυτή η συνεργατική οικονομία προσφέρει νέες ευκαιρίες, ανάπτυξη, απασχόληση, όμως ε, υπάρχει και ο κίνδυνος ε, να υπονομευτούν οι κοινωνικές, ε, τα κοινωνικά επιτεύγματα. Είπατε ότι θα συνεργαστείτε στενά και με τον υποψήφιο επίτροπο για την απασχόληση για να βρείτε ε, τις ε, σωστές ε, εργασιακές σχέσεις για όσους εργάζονται σε πλατφόρμες. Μπορείτε να μας πείτε πώς ακριβώς προβλέπετε να βελτιώσετε τη συνεργασία με άλλους επιτρόπους για να βελτιώσετε τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στις πλατφόρμες έτσι ώστε η οικονομία των πλατφορμών να είναι προστατευμένη μένει να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Κύριε Πρετών, πολύ σημαντικό ζήτημα. Ε, θα βρίσκεται στο επίκεντρο και των αλλαγών των ε, ανατροπών ε, στις οποίες αναφερόμαστε από την αρχή αυτής της ακρόασης και στο επίκεντρο φυσικά της στρατηγικής που αφορά το χαρτοφυλάκιο αυτό το οποίο ενδεχομένω θα μου αναθέσετε. Όλοι γνωρίζουν φυσικά ε, νέοι, λιγότερο νέοι που έχουν εργαστεί σε αυτέ τι πλατφόρμε, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των Ευρωπαίων έχουν κάποια στιγμή εργαστεί σε τέτοιε πλατφόρμε. και ξέρουμε πώ ε, αυτέ οι πλατφόρμε έχουν ένα χαρακτήρα κατάρριξη ουσιαστικά τη διαμεσολάβηση. Ε, έχουν δημιουργήσει οικονομικά μοντέλα απίστευτα. Δεν θα κάνω διαφήμιση τώρα για του μεν και του δε, αλλά όλοι γνωρίζετε σε τι αναφερόμαστε και ταυτόχρονα παρατηρούμε μια αβεβαιότητα Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Υπάρχει μια βεβαιότητα. Ε, κάνουμε λίγο λογοπαίγνια. Λέμε καταπληκτική. Αυτή η νέα γενιά είναι επιχειρηματίε μόνοι του. Αυτόνομοι και τελικά ανταποκρίνονται ε, στι φιλοδοξίε μα. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί νέοι σήμερα είναι επιχειρηματίε. Αυτό Αλλά αυτό δεν σημαίνει καταργούμε τα κοινωνικά δικαιώματα και εγώ ε, θέλω να εξετάσουμε ακριβώς αυτή την εξέλιξη και να επανέλθουμε ε, στα θεμέλια της κοινωνίας μας, να αρχίσουμε να δημιουργούμε υποχρέωσεις για το σύνολο αυτών των πλατφορμών και θα το κάνουμε βάσει συζητήσεων, συνομιλίων και αν αυτό δεν αρχίσει θα πάμε και πιο πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Βαν Σπάρεντακ, τη ΣΥΜΚΟ από τους Πρασίνους. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Η δημιουργία της κοινή αγοράς επέφερε ωφέλη στους πολίτες και στην οικονομία, αλλά όλο και περισσότερο βλέπουμε να υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα στη συνεχιζόμενη βάθυνση της κοινή αγοράς και στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πολίτη. Πρέπει να τους χάνει τομέα της υγείας. Εκεί υπάρχουν στην Ολλανδία τουλάχιστον πολύ αρνητικέ επιπτώσεις. Έχουμε ανθρώπους με ψυχιατρικά προβλήματα που κάθε μέρα τους φροντίζει κάποιος άλλος, δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό γιατί κέρδισε κάποιο άλλο τον διαγωνισμό. Πώ μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η ιστορική αγορά θα είναι ένα μοχλό έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και οι δημόσιε αρχέ να μπορούν να βελτιώνουν την κατάσταση και όχι να την παρεμποδίζουν, την ποιότητα κυρίω. Μετά την κατάσταση στην Ολλανδία, ε, ο πρώην Επίτροπος είπε ότι ε, υπάρχουν παραβιάσεις των ε, κανόνων της κοινή αγοράς, κυρίως αναφορά το θέμα του περιβάλλοντος και την έγκριση τύπου των αυτοκινήτων. Αλλά η ποιότητα της ατμόσφαιρας ε, δεν αφορά μόνο τα αστικά κέντρα. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσον πραγματικά θα μπορέσετε να ελέγχετε τους, τις, τα αυτοκίνητα με μηχανές εσωτερικής καύσης. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Το πρώτο σας ερώτημα έχει να κάνει περισσότερο με την ελπίζω μελλοντική συναδελφό μου, την κυρία Κυριακίδη, γιατί εκείνη είναι υπεύθυνη για τα θέματα υγείας. Έχω ένα αρκετά ευρύ χαρτοφυλάκιο, δεν θα προσθέσω για την υγεία, παρόλο, παρόλο που τα θέματα της υγείας συνδέονται με τις υπηρεσίες και με άλλα. Αλλά είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό και η κυρία Κυριακίδου είναι εκείνη που θα το εξετάσει υπό την οπτική γωνία που λέτε. Εγώ θα σταθώ δίπλα της φυσικά, αλλά εκείνη μπορεί να απαντήσει στο ερώτημά σας. Το δεύτερο τώρα. Ε, το συνδυάζω με το Dieselgate, φαντάζομαι αυτό έχετε κατά νου. Με τις συνέπειές του και με την ουδετερότητα απέναντι στον άνθρακα που θέλουμε να έχουμε το 2050. Μη φοβόμαστε τις λέξεις. Το Dieselgate ήταν ένα σκάνδαλο. Και χάρη στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και εδώ χαιρετίζω το έργο της ε, Εξεταστικής Επιτροπής εδώ, κατέδειξε τι συνέβη. Τώρα, για να απαντήσουμε στο σκάνδαλο αυτό, κάποιες χώρες αρχίζουν να θέτουν προδιαγραφές, αλλά υπάρχει και το ζήτημα που έχει να κάνει με το οχήματα μηδενικών εκπομπών. Κάποιες χώρες το συζητάνε, όπως επίσης και κάποιοι κατασκευαστές. Το βρίσκω καλό. Δεν λέω ότι υπάρχει μόνο αυτό, αλλά ναι. Και τοπικά υπάρχουν κίνητρα με χρηματοδότηση. Πρέπει να τα ενθαρρύνουμε, ναι, αλλά να μην αποσταθεροποιηθεί η εσωτερική αγορά. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Πάντως, ε, κατόπιν τη συνειδητοποίηση και οι χώρες αρχίζουν να επιταχύνουν την προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Υπήρου προς την κατεύθυνση της ουδετερότητας στον άνθρακα που θέλουμε να έχουμε το 2050. Αρκεί να είμαστε πάντα συμβατοί με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Σαφώς και είμαι υπέρ. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. ευχαριστώ για την απάντησή Σε Ορισμένα πράγματα δεν τα κατάλαβα καλά. Εξακολουθώ να μην τα έχω καταλάβει, γιατί κατ' ουσίαν μιλάμε για την υγεία των πολιτών μα, για την ποιότητα ε, τη ατμόσφαιρας, για τον αέρα που αναπνέουμε όλοι μα ε, και είναι κακής ποιότητα αυτό ο αέρα. Ε, ένα βασικό αίτιο είναι οι μηχανέ εσωτερική καύσης. Πιστεύετε ότι η κοινή αγορά θα πρέπει να υπερέχει των φιλοδοξιών μα για την κλιματική αλλαγή και τι ποιότητας της ατμόσφαιρας, της ποιότητας του αέρα. Μανέκια, ναι, και πάλι λέω ότι η φιλοδοξία μας, πώς συλλογικά την αποφασίσαμε με την εκλεγμένη πρόεδρο Φοντερ Λάιεν, να πετύχουμε μηδανικέ εκπομπές άνθρακα, είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει, να επιταχύνουμε. Συμφωνώ μαζί σας, ο αέρας που αναπνέουμε θα επηρεαστεί, ευτυχώς, από τις αποφάσεις μας. Οπότε θα ενθαρρύνω να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και μάλιστα προς την κατεύθυνση που είπατε κι εσείς. Και κατά τα άλλα, επειδή πριν μίλησε για το Dieselgate, να λάβουμε υπόψη μας και την συμμόρφωση των οχημάτων. Γιατί η πιστοποίηση αυτή της συμμόρφωσης χρησιμοποιείται από κάποιου για να πούνε ότι γι' αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά δεν ισχύει αυτό. Η Κίνα τα χρησιμοποιεί. Εμείς Πώς είμαστε στα 60, θέλουμε να πάμε στο 80, οπότε κάποιες ήπειροι προχωράνε προς την κατεύθυνση που είπατε. Οπότε και εμείς, ναι, θέλουμε να γίνουν οι προσαρμογές αυτές ε, στη βιομηχανία, στον κλάδο. Αλλά είναι το όραμα, βλέπετε, του Αντιπροέδρου Τίμερμαν που θα οδηγήσει και τους άλλους να πάνε προς την κατεύθυνση που εσείς λέτε. Ευχαριστούμε. Επόμενη μιλήτρια είναι η κυρία Ίσκρα Μιχαλάγιοβα. Ήτρε από τη Ρινιού. Παρακαλώ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, κύριε υποψήφιε Επίτροπε, το μελλοντικό σας χαρτοφυλάκιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία ε, στις ε, προοπτικές ε, της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, στην ανταγωνιστικότητά της και στην εξέλιξή της μέσα από τον αυτοματισμό και την ψηφία η ανταγωνιστική βιώσιμη ευρωπαϊκή βιομηχανία συνεπάγεται πάρα πολλά ωφέλη στην κοινωνία και στην οικονομία μας. Παρ' όλα αυτά έχουμε βιομηχανικούς τομείς όπως ο τομέας των κατασκευών όπου ε, δεν υπάρχει ουσιαστικά ψηφιοποίηση και ρωτώ εσείς ε, πώς ακριβώς ε, μπορείτε να διασφαλίσετε μεγαλύτερη ψηφιοποίηση στον τομέα των κατασκευών και σε γενικές γραμμές πώς μπορείτε να δώσετε κίνητρα για να επεκταθούν τα ψηφιακά επαγγέλματα και η ψηφιοποίηση γενικότερα σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, το είπα και προηγουμένως. Όλοι οι τομείς της εσωτερικής αγοράς χαρακτηρίζονται από την ψηφιοποίηση. Και συμπεριλαμβανομένου, και ευχαριστώ που το θυμήσατε γιατί μερικές φορές το ξεχνάμε, ο βασικότατος τομέας της οικοδομής. Το 9% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Υπενθυμίζω 3 εκατομμύρια επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είναι τεράστιο. Και εκεί ωστόσο παρατηρώ τις ανατροπές, ε, ε, τις ψηφιακές που θα είναι σημαντικότατες. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα, την κατασκευή συγκεκριμένων ε, εξαρτημάτων με εκτύπωτες τρισδιάστατης εκτύπωσης. Πρέπει να είναι κανείς και μηχανικός και πληροφορικάριο. Είναι διπλή η μόρφωση που χρειάζεται. Όλα όσα αφορούν επίση τη χρήση ιδιαίτερων τεχνολογιών ε, και ειδικότερα να επανέλθουμε σε αυτούς που υπερασπίζονται όπως και εμένα τα διαφορετικά τα δεδομένα, τεχνολογίες σημαντικές, αισθητήρε, οπτικοί που μετρούν με ακρίβεια χιλιοστού κινήσεις, ε, στηρίξεις ε, που έχουν ένα όραμα ε, δίνουν εικόνε των πάντων, των υπογείων. Όλο ο τομέα των οικοδομών λοιπόν χαρακτηρίζεται από άκρη σ' άκρη από την ψηφιακή τεχνολογία. Οπότε, ε, όπως είπα, θα χρειαστεί ε, κατάρτιση επιτόπου σε πραγματικέ συνθήκε για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε αυτέ τι τρει εκατομμύρια επιχείρησει που πολλέ από αυτέ είναι μικρομεσαίες. Ε, να επανεκπαίδευση λοιπόν στι ψηφιακές καινοτομίε, ώστε αυτέ οι κατασκευαστικέ επιχειρήσει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία ψηφιακά, ψηφιακά ανάλυση δεδομένων, ε, τεχνητής νοημοσύνης που θα αναπτυχθούν στον κλάδο. Το πρόγραμμα λοιπόν όλα αυτά ε, που θα ε, υποστηρίξει ε, ψηφιακού πόλου ενημέρωση, θα βοηθήσει ε, την οικοδομή διαθέτοντας στον ευρωπαϊκό χώρο όλες τις σχετικές πληροφορίες. Ευχαριστούμε. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Σας ευχαριστώ ε, για την πολύ συγκεκριμένη και εμπεριστατωμένη απάντησή σας. Ε, τώρα, συμπληρωματική ερώτηση. Στο χαρτοφυλάκιό σας... Έχετε την ψηφιοποίηση της Ευρώπης. Ένα κριτήριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανία προχωρούν χέρι-χέρι. Μήπως μπορείτε να μας ε, μιλήσετε λίγο περισσότερο για το όραμά σας, ε, για την ευρωπαϊκή στρατηγική και για την ε, στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Ρεμπερτό. Πέντε είναι τα βασικά σημεία του προγράμματος αυτού. Πέντε σημεία που οριοθετούνται, τα έχουμε πει καθαρά, τα επαναλαμβάνω γιατί είναι σημαντικά για μένα. Τα κανονιστικά και διοικητικά εμπόδια είναι το πρώτο. Δεύτερον, βελτίωση Τη εφαρμογή τη οδηγία για τι ε, καθυστερήσει πληρωμών. Ε, σε αυτό οφείλεται το 30% των χρεοκοπιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τρίτον, υποστήριξη τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί έχουμε εργαλεία, θα την αυξήσουμε. Τέταρτον, προσαρμογή, το είπαμε προηγουμένω, ε, σε ενιαία αγορά στι ιδιαιτερότητε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να άρουμε τα σημεία συμφόρηση. Και πέμπτον, ανάπτυξη ικανοτήτων και ειδικότερα σε ψηφιακά θέματα. Το είπα και είναι πολύ σημαντικό και δεν το είπα προηγουμένω, αλλά είναι πολύ σημαντικό για την ε, βιωσιμότητα, γιατί όταν μιλάμε για κτίρια αναφερόμαστε στη ξεμόναση, ε, κτίρια μηδενική κατανάλωση ενέργεια, μηδενικών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Είναι σημαντικά θέματα. το έχω συζητήσει με τον Επίτροπο Νικολάη Σμιτ, οπότε θα συνεργαστούμε προφανώ και αυτό το τελευταίο σημείο. Το επαναλαμβάνω, είναι σημαντικό θέμα ε, ο εντεταλμένο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που δεν έχω ορίσει ακόμα, φυσικά δεν έχω ορίσει κανέναν ακόμα, είναι πρόωρο, θα παίξει σημαντικότατο ρόλο ω ε, ε, εκπρόσωπο τη Κομισιόν το για τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Έιλερ. Παρακαλώ. Ε, σύντομη θα είναι η ερώτησή μου, κύριε υποψήφιε επίτροπε, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που προκύπτουν όταν οι οικονομίες όπως η Κίνα αγοράζουν την τεχνολογία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Μπρετό. Θα απαντήσω με μια απάντηση λίγο μεγαλύτερη από την ερώτηση που κάνατε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό, πολύ ευρύ. Πρώτα απ' όλα, να υπενθυμίσω, η πρώτη ερώτηση είναι θέμα κυριαρχία και ηγεσία στον τεχνολογικό κλάδο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον κόσμο να κάνει την άνε. και στη δική σα χώρα, στη Γερμανία, κύριε Έλερ, είδαμε τελευταία ότι κάποια πράγματα ίσω να μην έπρεπε να είχαν γίνει. Ε, θα έπρεπε να έχει δοθεί λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Αναφέρθηκα σε αυτά τα πράγματα. Οπότε α μην είμαστε αφελεί. Α μην είμαστε αφελεί. Πρέπει να ξαναδούμε, όπω είπα προηγουμένω, δεδομένων των όσων συμβαίνουν ε, στι χώρε μα και γύρω μα ε, θα πρέπει να ξαναδούμε, να αναθεωρήσουμε τι πολιτικέ που θα επιτρέψουν να προστατευτούμε στο πλαίσιο των κανόνων της αγοράς. Α θυμηθούμε του κανόνες οδηγία οδηγίας ε, για τι υπηρεσίε, Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και πολύ περισσότερο τα εργαλεία φιλτραρίσματος των άμεσων επενδύσεων για να ε, προστατεύσουμε την τεχνολογική μας ε, κυριαρχία, όπως κάνουν και άλλε ήπειροι. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη διανοητική ιδιοκτησία με στόχο την τεχνολογική ε, κυριαρχία, ηγεσία. Δεν συμβαίνει ακόμα αυτό, την τεχνολογική μας ανεξαρτησία. Θα πρέπει επίσης να αναπτύξουμε σε αυτούς τους κλάδους μια πολιτική αλυσίδα παραγωγή ε, ουσιαστικά σχέδια κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντο που θα μα επιτρέπουν, όπω αυτό για τι μπαταρίε, ε, που θα μα επιτρέπουν να έχουμε παρεμβάσει μαζικέ, να επανακαθορίσουμε ολόκληρε αλυσίδε παραγωγή και να επανοικοδομήσουμε σημαντικά κομμάτια τη βιομηχανία ε, στα οποία Δυστυχώ δεν είχαμε προχωρήσει επαρκώ, ενώ άλλε υπήροι που δεν είχαν τα ίδια προληπτικά μέτρα είχαν χρηματοδοτήσει επιχειρήσει. Ε, και έτσι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε και εμεί επιχειρήσει που θα έρχονται στην επικράτειά μα. Ευχαριστώ. Ε, Συμπληρωματικέ ερωτήσει. Στην πολιτική όπω και στη ζωή, μερικέ φορέ η δεύτερη αγάπη μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή για γάμο. Ακούσαμε προσεκτικά όταν δεσμευτήκατε να τηρείτε τον κώδικα διοντολογία τη Κομισιόν που διασφαλίζει ότι ότι ο λομπίστα δεν είναι πια λομπίστα όταν γίνεται επίτροπο, ότι ο επιχειρηματία δεν είναι πια λομπίστα για την επιχείρησή του, ότι ένα Γάλλο επίτροπο θα δρά για όλου του Ευρωπαίου. Αυτό που ακούσαμε σήμερα ουσιαστικά αποτελεί διακριτική μεταχείριση προ ανθρώπου που είχαν επιτυχία στον οικονομικό κλάδο. Θεωρείτε ότι θα καταφέρετε να είστε επιτυχεί ω ε, επίτροπος. Αυτή είναι η δεύτερη μου ερώτηση. Και τώρα ο κύριος Επίτροπος, ο Επιστήφης Επίτροπος έχει πέντε λεπτά για να κλείσει την παρουσίασή του. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταλλαγή που είχαμε. Πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάστηκα για να ετοιμάσω, να ετοιμαστώ για τις απαντήσεις σας, κάπως πρωτότυπος. Είχα τους συνεργάτες μου, οι οποίοι με προετοίμασαν σε πολύ λίγες μέρες, γιατί είχα λίγο χρόνο. Λοιπόν, αντί να περάσω το χρόνο μου με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ένα τέταρτο πέρασα με το Γενικό Διευθυντή της Connect και άλλο τόσο με την Growth, αλλά προσπάθησα αυτές τις μέρες να δω όσο γίνεται περισσότερους από εσά. Δεν μπόρεσα να σας δω όλου βέβαια, αλλά κάπου 50 είδα. Και αυτό με προετοίμασε. Γιατί εσείς είσαστε οι πολιτικοί που θέλω να υλοποιήσω. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι απόφαση και αν πάρετε είναι μια υπέροχη ανθρώπινη περιπέτεια και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Αν αποφασίσετε ότι είμαι ο κατάλληλος, αυτό θα αποτελέσει και τη βάση για τις ε, υπόλοιπες σχέσεις μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις τρεις προκλήσεις της Ευρώπης στο γεωπολιτικό πλαίσιο που βρισκόμαστε. Εγώ το λέω, το επαναλαμβάνω, έχουμε το περιβάλλον, τα ψηφιακά και το κοινωνικό. Αυτές είναι οι τρεις προκλήσεις μας. Και για να δώσουμε απάντηση σε αυτές, εγώ τουλάχιστον θα χρησιμοποιήσω όλη την ενέργεια που διαθέτω για να προστατεύσουμε καλύτερα την εσωτερική αγορά, να βοηθήσουμε στην ε, τροποποίησή της και η πυρός μας έτσι να γραφεί στον 21ο αιώνα πραγματικά. Δεν έχουμε χρόνο όμως, επήγει η κατάσταση. Η κατάσταση δεν είναι αυτή που θα θέλαμε, αρκεί να δούμε τι γίνεται στους διάφορους αυτούς κλάδους για να καταλάβουμε ότι σε όλους αυτούς πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα, βάσει των αξιών μας. Δεν έχουμε απελευθερώσει το δυναμισμό που έχουμε στη διάθεσή μας, ούτε στον ψηφιακό τομέα, ούτε αλλού. Αλλά είναι απ' την άλλη εξαιρετικό νέο, γιατί σημαίνει ότι εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε στη διάθεσή μας πόρους που δεν έχουμε ακόμα εκμεταλλευτεί. Και εμείς οι ίδιοι ε, μερικές φορές εμποδιζόμαστε από κάποιες προσεγγίσεις ξεπερασμένες. Συνεπώς η Ευρώπη μας πρέπει και μπορεί να αποτελέσει το οικοσύστημα του 21ου αιώνα που να διαρθρώνεται γύρω από τις τρεις προκλήσεις που σας είπα πριν. Ένα οικοσύστημα και υπηρεσίες προς όλους, προς όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους συμπολίτε μας με τη δικιά σας εμπιστοσύνη ε, θα ε, χρησιμοποιήσω όλη μου την ενέργεια τα επόμενα πέντε χρόνια ε, μαζί σας, στο πλευρό σας. Αν με εμπιστευτείτε και μου επιτρέψετε να συνεχίσω στο δρόμο που πάντα ακολουθούσα, πάντα επικοδομητικά θα δουλεύω. Η διακυβέρνηση είναι κάτι που έχω στην καρδιά μου. Ξέρω ποιοι είσαστε, εσείς εκπροσωπείτε τους λόγους της Ευρώπης, οπότε θα συνεργαστούμε ο καθένας από την θέση του την ανεξαρτησία πνεύματός μου επίσης. Ελπίζω να το αισθανθήκατε αυτό. Ε, θα την βάλω στην υπηρεσία του κοινού μας σκοπού ε, για το επιχειρίζεστε, τη διακυβέρνηση υπέρ της Ευρώπης μας. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει το νήμα της ιστορίας της. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από μία ενια αγορά είναι μία κοινότητα, μία κοινότητα αλληλεγγύης, συγκλήσεων, σεβόμενη τις διαφορές και υπέρ της ενότητας για να βαραίνει στον κόσμο. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ό,τι μέσα διαθέτω, όλη μου τη δύναμη και την έργεια. Και το καταλάβατε, δεν είμαι και αφελής από την άλλη. Ξέρω αυτά που μου έμαθε η ζωή. Η πρόοδος οδηγεί στην πρόοδο, η επιτυχία οδηγεί στην επιτυχία. Και αυτά θα τα πετύχουμε εφόσον συνεργαστούμε χέρι-χέρι με εσά, τους εκπροσώπους των 500 εκατομμυρίων ε, ανθρώπων της Επίρου μας, βάσει των αξιών μας, της ελευθερίας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, Συνάδελφοι, σας αγαπώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Και ευχαριστούμε κύριε υποψήφιε επίτροπε για τις απαντήσεις σας, για αυτά που μας είπατε στο τέλος. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σούτερ, Σούτερ, για να κλείσει τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τις δύο επιτροπές, τον υποψήφιο επίτροπο. Ευχαριστώ και όλους όσοι συνέβαλαν στην οργάνωση αυτής της συνάντησης, στη γραμματεία. Ε, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά για να ετοιμάσουμε αυτή τη συνεδρία. ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει Πρόεδρος. Θα βρεθούμε σύντομα για να αποφασίσουμε σε σχέση με την ακρόαση αυτή. Θα δώσω στον κύριο Γρασνοδεύσκη το λόγο για να κλείσει αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θέλω να ανακοινώσω ότι και κλεισμένων των θυρών στις 5 εδώ θα συνεδριάσουν οι συντονιστές από τις δύο επιτροπές για να αποφασίσουν για την ακρόαση αυτή. Ευχαριστώ.